that you can directly go to. Okay, so good morning everyone. Sorry for being a few minutes late. We will start with... Καλημέρα σε όλους. Ε, συγγνώμη που έχουμε καθυστερήσει λίγο. Θα ξεκινήσουμε με την εξέταση των τροπολογιών για το σημείο 6 της ημερησίας διάταξης. Ναι, ο εισηγητής, έχετε δίκιο, δεν είναι εδώ, αλλά εγώ θα κάνω μια δήλωση εκ μέρους του. Προεδρεύω και με εισηγητής. Ε, έχουμε χρόνο μέχρι τις 9.30 όπου θα έρθει ο κύριος Αλμούνια, γι' αυτό θέλω να ξεκινήσουμε γρήγορα. Σημείο 6. Προσχώρηση της Κροατίας στη σύμβαση της 23ης Ιουλίου 1990 για την εξάλληψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Ο εισηγητής κύριος Νίτρας του ΕΛΚ δεν καταφέρει να φτάσει στις Βρυξέλλες λόγω καθυστέρησης του αεροσκάφους. Έτσι, εκ μέρους του θα ανακοινώσω εγώ μια δήλωση. Η έκθεση αφορά την προσχώρηση της Κροατίας ε, στη συνθήκη που αποσκοπεί στην εξάρτηση της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεων των κερδών συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Ο κανόνα του Κοινοβουλίου σε αυτή τη διαδικασία είναι να κάνει μια σύσταση υπό τη διαδικασία διαβούλευσης. Πιστεύουμε ότι αυτός ο φάκελος δεν θα παρουσιάσει προβλήματα, κανένας και ο δεν εξέφρασε επιφυλάξεις και δεν υπάρχει πρόβλημα με την προσχώρηση της Κροατίας στη συνθήκη αυτή με εφαρμογή των σχετικών μέσων ε, στις συντομότερες προθεσμίες. Έχουν ε, συμφωνήσει σκιώδεις για το σχέδιο. Υπάρχει μία τροπολογία του κ. Μπρουσατομάσικ του ECR. Υπεογράμισε την ανάγκη να τεθεί σε ε, εφαρμογή το ταχύτερο η συνθήκη αυτή ώστε να ελαφρύνει το φόρτο των, ε, της Κροατίας ε, των κρατών επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στην εσωτερική αγορά. Κάτι πολύ επωφελές. Ε, πολύ επωφελής αυτή η τροπολογία θεωρείται από τον εισηγητή και θα ληφθεί υπόψη. Ο εισηγητής προτείνει να προχωρήσουμε και να ψηφίσουμε την έκθεση σήμερα την απογευματινή συνεδρίαση. Κύριε Λούδιξον. ο κύριος Λούδιξον δεν είναι εδώ. Δεν ξέρω αν κάποιος θα ήθελε να πάρει τον λόγο εκ μέρους του κύριου Λούδιξον. αλλιώς ο κύριος Τρεμόσα. Ε, ευχαριστώ. Πρόεδρε. Είναι τεχνικό το θέμα αυτό. Ε, δεν έχει κάποιο μακρό ιστορικό. Όσοι φιλελεύθεροι θα ε, ψηφίσουμε υπέρ βοηθάει την Κροατία να γίνει ένα κανονικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ό,τι αφορά αυτή την τροπολογία, όπως είπατε υπάρχει μόνο μία τροπολογία που έχει κατατεθεί, μπορούμε να σκεφτούμε ότι το θέμα αυτό είναι τεχνικό και η τροπολογία αυτή είναι πιο πολύ ιδεολογική διότι υπογραμμίζει την ανάγκη να μειωθεί το φορολογικό άχθος ε, επί των φορολογουμένων ως μεσογειακός ε, εκπρόσωπος χώρας Μεσογείου ε, συμφωνώ με την τροπολογία αυτή θα συζητήσω και με τα άλλα μέλη της ομάδας και θα δούμε από την άλλη μεριά αν ο εισηγητής συμφωνεί εξασφαλίζεται πλειοψηφία μεταξύ του ΕΛΚ, του ΙΣΙΑΡ και των άλλων ενδεχομένων ομάδων θα δούμε χτες την ομάδα, στην συνάντηση ομάδα των φιλελευθέρων ε, διερωτώμασταν αν τέτοιου είδου πολιτικέ τροπολογίε πρέπει να μπαίνουν σε, τεχνικά, σε τεχνικές εκθέσεις. Εγώ δεν έχω πρόβλημα προσωπικά, αλλά κάποιοι άλλοι συνάδελφοι μπορεί να διαφωνούν, οπότε θα το δω με του συναδέλφου. Δεν ήξερα ότι το ΕΛΚ υποστηρίζει αυτή την τροπολογία και δεν ήξερα καν ότι το, οι Ευρωπαίοι συντηρητικοί μεταρρυθμιστές την είχαν καταθέσει. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Θέλει κανείς άλλο το λόγο. Κύριε Μάλετικ. Ως Ευρωβουλευτής από την Κροατία θα ήθελα να καλημερίσω όλους τις, τους συναδέλφους και να ευχαριστήσω όσους εργάστηκαν πάνω στην έκθεση αυτή, ιδιαίτερα τον εισηγητή τον κύριο Νίτρας θα ήθελα να πω ότι η τροπολογία της κυρίας ε, Τόμασης αποτελεί μια σημαντική δήλωση μέσα στην έκθεση αυτή και πιστεύω ότι μπορεί να γίνει αποδεκτή διότι αποτελεί σημαντικό μέρος ε, της ε, πλήρους ένταξης της Κροατίας στην ενιαία αγορά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την επιχειρηματική μας κοινότητα. Ευχαριστώ. Θα ψηφίσουμε λοιπόν σήμερα πάνω στην έκθεση και θα πάει στην Ολομέλεια, στην δεύτερη Ολομέλεια του Απριλίου. Περνάμε στο επόμενο θέμα της ημερησίας διάταξης, ε, το σημείο 7, κοινό φορολογικό καθεστώς, το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις ε, θηγατρικές εταιρείες ε, διαφορετικών κρατών μελών. Η συγγήτρια είναι η κυρία Κλέβα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω όλου του σκιώδη εισηγητές και άλλου συναδέρφους που υπέβαλαν τροπολογίε πάνω στην έκθεσή μου. Εξετάζουμε μικρό αριθμό τροπολογιών που στις περισσότερες ε, περιπτώσεις είναι είτε συμπληρωματικές σε σχέση με τη δική μου διατύπωση ή είναι κατά. Ε, φαντάζομαι ότι όλοι θα συμφωνήσετε ότι ε, δεν είναι απαραίτητο να γίνουν επιπλέον συμβιβασμοί στις περιπτώσεις αυτές κάποιες γενικές παρατηρήσεις ε, για το θέμα αυτό. Χαίρομαι πάρα πολύ που η Κομισιόν ε, με αυτή την επικαιροποίηση ε, τις οδηγίε για τι μητρικέ και τι θηγατρικές εισήγαγε δύο τροποποίησει που ζητάει εδώ και πολύ καιρό το Κοινοβούλιο. Το θέμα των υβριδικών δυσαναλογιών, των υβριδικών ασυμφωνιών και τον κανόνα για τον, για τον Γενικό Κανόνα Απαγόρευση Καταχρήσεων. Και, Πιστεύουμε ότι το θέμα αυτό θα πρέπει να το χειριστούμε πολύ γρήγορα. Είναι κάτι το οποίο έχουμε ζητήσει επανειλημμένα. Ε, εδώ και το ίδιο ισχύει και για τον κανόνα περί καταχρήσεων. Ε, ε, και πιστεύω ότι έτσι βάζουμε τέλος στην στο ε, αρμπιτράζ ε, όπου οι επιχειρήσεις ε, προσπαθούν να αναζητήσουν τα πιο ευνοϊκά καθεστώτα. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε τέλος στα φορολογικά ωφέλη που προκύπτουν από την ελληπή ρύθμιση. Χαίρομαι πολύ που περισσότεροι ευρωβουλευτές συμφωνούν με τις διατάξεις που εμποδίζουν περαιτέρω στρέβλωση της ανταγωνιστικότητας. Ε, πάντα ήμουν υπέρ της θέσης ε, του Κοινοβουλίου απέναντι στο CCTV, αλλά επειδή είχε παγώσει το θέμα αυτό στο Συμβούλιο, πιστεύω ότι πρέπει ε, να κάνουμε περισσότερα όσον αφορά τους συντελεστές φορολογίας εταιριών στις χώρες μας. Προτείνουμε ο συντελεστής αυτός να μην είναι χαμηλότερος από το 75% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, υπολογίσαμε ότι έτσι καταλήγουμε σε συντελεστή 15,5%. Ε, κάτι που σημαίνει ότι οι πέντε κράτη-μέλη θα βρίσκονται κάτω από το κατόφλι. Πιστεύουμε ότι οι συντελεστές φορολογίας μπορούν να λειτουργήσουν καλύτερα και το να συγκρίνουμε τον πραγματικό συντελεστή φορολογία αυτή τη στιγμή είναι πολύ πιο δύσκολο από το να συγκρίνουμε του νόμου συντελεστέ φορολογία εταιριών. Ο συνάδελφο Κίκολ δυστυχώ δεν είναι παρόν σήμερα, αλλά εισήγα και παρόμοιε τροποποιήσει στην ε, δική του έκθεση πάνω στην οδηγία του 2011 και ελπίζω να στηρίξετε τις τροπολογίες αυτές. Είναι η τελευταία μου έκθεση αυτή και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις εισηγητές για την επικοδομητική συνεργασία που είχαμε τις περασμένες εβδομάδες. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Κλίβα. Ο κύριος Κλίντς έχει ζητήσει το λόγο. Βάλτε τα ακουστικά να μιλήσω γερμανικά, παρακαλώ. Also grundsätzlich, ε, Κατά βάση, πρέπει να επικροτήσουμε την πρόταση αυτή που στόχο έχει την... να δώσει τέλος στην φοροαποφυγή. Έχω όμως ε, μία παρατήρηση όσον αφορά την τεχνική εφαρμογή της πρότασης. Η εισηγήτρια έκανε μία πρόταση Ε, στο κράτος ε, μέλος ε, αποδοχής να υπάρχει φοροπαλλαγή εάν στο κράτος μέλος προέλευσης πληρώνεται φόρος με νόμιση τελισή το 75% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Αυτό στην πράξη όμως είναι δύσκολο να γίνει, διότι είναι δύσκολο να υπάρξει σύγκριση των, νομίμων συντελεστών, διότι μπορεί μια χώρα με υψηλότερο νομικό, νόμιμο συντελεστή να είναι πιο ελκυστική, επειδή μπορεί να υπάρχουν άλλα πλεονεκτήματα. Μπορεί να υπάρχουν εξαιρέσεις, ενώ μια χώρα με χαμηλότερο συντελεστή φορολογίας ε, να μην επιτρέπει εξαιρέσεις. Έτσι λοιπόν Θέλουμε να αποφύγουμε τη διπλή φορολόγηση, αλλά στην πράξη μπορεί τελικά στο κράτος μέλος προέλευσης και στο κράτος μέλος ε, αποδοχής τελικά να έχουμε ε, μη φορολόγηση κάτι που δεν είναι στο πνεύμα του κειμένου. Όταν μιλάμε για φορολογία εταιριών, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ε, χώρες που πέρα από αυτόν ε, τον φόρο έχουν ένα επιπλέον φόρο, κάτι που ισχύει στη Γερμανία, ε, όπου υπάρχει φόρος άσκησης επαγγέλματος και γι' αυτό στις τροπολογίες 10 και 11 Έχω αμφιβολίες εάν είναι σκόπιμα αυτά που αναφέρονται. Ευχαριστώ. Ωραία, ο κύριο Κλίντ, κύριε Στολόγιαν, θέλετε το λόγο. Ναι, ευχαριστώ. Είχαμε μια εξαιρετική συζήτηση στην πολιτική μας ε, ομάδα όσον αφορά την έκθεση αυτή. Υποστηρίξαμε διάφορες ε, τροπολογίες. Σύμφωνα με τον κύριο Κλίντ. Δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε τις τροπολογίες που υποτίθεται ότι ορίζουν τέτοια όρια όπως για παράδειγμα συντελεστή εταιρικής φορολόγησης όχι χαμηλότερο από το 75% του ε, νόμιμου φόρου που προβλέπεται δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε τέτοιου είδους ε, κατόφλια διότι πρώτα απ' όλα έχουμε χώρες όπου η φορολογική πολιτική είναι σαφής και αποτελεί θέμα εθνικής πολιτικής και όχι ευρωπαϊκής. Επίσης υπάρχει άλλη μια τροπολογία προφέρω το 10% συμμετοχή στο κεφάλαιο μιας εταιρείας και η πρόταση είναι να αυξηθεί σε 15%. Εμείς θεωρούμε το 10% είναι μια χαρά. Κατά τα άλλα υποστηρίζουμε την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ. Ωραία, ευχαριστούμε κύριε Στρόιαν. Δεν ξέρω αν η Κομισιόν θα ήθελε να πάρει το λόγο. Όχι, όπως βλέπω. Θα δώσω ξανά το λόγο λοιπόν στην κυρία Κλέβα. Ναι, θα συμφωνήσω. Όπως είπαμε στην αρχή στις τροπολογίες υπήρχαν δύο επιλογές μόνο, υπέρ ή εντελώς κατά ε, της πρότασής μου. είναι μακρά ιστορία της υπόθεσης αυτής. Πιστεύω, ελπίζω ότι μια μέρα θα έχουμε εναρμόνιση φορολογική στην Ευρώπη. Και αυτό το θέμα οδηγεί σε διχονομία μεταξύ των διαφορών πολιτικών ομάδων. Βλέπω ότι ο καθένας ε, έχει διαφορετικές θέσεις. Συμφωνώ επίσης. Είναι πολύ δύσκολο να συγκρίνουμε τους διάφορους συντελεστές φορολόγησης στα διάφορα κράτη-μέλη. Σίγουρα ήταν ε, και δύσκολος αυτός ο υπολογισμός του 15,5% αλλά κάναμε ότι μπορούσαμε καλύτερο. Ε, ίσως ε, προσπαθήσαμε να είμαστε λίγα πιο φιλόδοξοι ώστε το νέο κοινοβούλιο να έχει περισσότερες δυνατότητες διαπραγμάτευσης. Όπως είπα στην αρχή, οι ενοιολογικές διαφορές ήταν σαφές μετά από την κατάθεση των τροπολογιών. Ας πάμε στην ψηφοφορία και θα δούμε τι θα συμβεί. Ευχαριστώ πολύ κυρία Κλέβα. Θα ψηφίσουμε σήμερα για την εκθέση αυτή. Θα ψηφιστεί, υποψηφιζόμαστε στην επόμενη Ολομέλεια του Απριλίου. Θα διακόψουμε για λίγα λεπτά μέχρι να ξεκινήσουμε το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη, την ανταλλαγή απόψεων με τον Επίτροπο κ. Αλμούνια. Αναμένουμε λοιπόν την αύξησή του. Και κάνουμε μια διακοπή πέντε λεπτά. Ευχαριστώ. Okay, um, we may resume now. Uh, Συνεχίζουμε τώρα τη συνεδρίασή μας με μεγάλη χαρά. Καλώς ορίζω τον Επιτρόπο κ. Αλμούνια σε αυτή την τελευταία ανταλλαγή απόψεων. Ζητώ συγγνώμη. Α, να, δεν θα μπορώ να μιλήσω κάποια στιγμή, έχω βροχίτιδα. Γι' αυτό είπα στον κύριο Επίτροπο ότι δεν μπορεί να μου δώσει ένα φιλί. Δεν έχει να κάνει με αυτόν. Απλά σε περίπτωση που αυτό ε, προβληθεί live ε, στο web stream, ε, να μην νομίζει κανείς ότι δεν συμπαθώ τον κύριο Επίτροπο. Είναι η τελευταία φορά που βρίσκεται μαζί μας στην ΕΚΟΝ ο κύριος Αλμόνια και θα ήθελα να τον καλωσορίσω και να τον ευχαριστήσω για την εξαιρετική συνεργασία του με το Κοινοβούλιο και ειδικότερα με την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας. Έχουμε ακούσει κάποιες πληροφορίες για το ποια θα είναι η στάση σας ε, όταν ακούσαμε την ακρόαση σας ως Επιτρόπου και έχω εδώ τρεις ερωτήσεις για εσάς. Ε, πώς θα συνεργαστείτε με το Κοινοβούλιο και είπατε ότι ναι, θα συνεργαστείτε και προσφερθήκατε να υπογράψετε αυτή την υπόσχεση και αυτό δημιουργεί έτσι μια τάση γιατί να ζητήσουμε τέτοιες υποσχέσεις από όλους τους επιτρόπους. Ε, σε ζήτησα να στείλετε ένα έγγραφο σε πρώιμο στάδιο ώστε η λήψη αποφάσεων στην Κομισιόν ε, στον τομέα του ανταγωνισμού να είναι αποτελεσματική και σε ζητάμε συνεργασία και ε, υποβολή αναφορών ε, σε όλα τα χαρτοφυλάκια οικονομικών θεμάτων. Δεν ήσασταν τέλειος, αλλά έχετε κάνει αρκετά καλή δουλειά και έχουμε προοδεύσει αρκετά στη διάρκεια αυτής της θητείας. Ελπίζω λοιπόν ότι ο νέος Επίτροπος και η νέα Επιτροπή ΕΚΟΝ θα συνεχίσουν αυτές τις εξαίρετες πρακτικές που ξεκινήσαμε εμείς. Ελπίζουμε ότι θα καθιερωθεί και ένας πλήρης ε, διάλογος περί ανταγωνισμού, όπως αναφέρουμε και σε μια έκθεση. Αυτή η συνεργασία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει πολιτικό διάλογο και λογοδοσία αφενός, καθώς και έγκαιρη ανταλλαγή πληροφορίων από την άλλη ώστε να συνεχίσουμε με βάση τα όσα έχουμε επιτύχει μέχρι τώρα. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που βρισκόσταν εδώ στην Επιτροπή ΕΚΟΝ όποτε το ζητήσαμε. Μάλιστα εσείς ζητήσατε να είστε πιο συχνά ακόμα και εμείς δεν είχαμε αρκετό χρόνο γι' αυτό λόγω του υψηλού φόρτου που είχαμε όσον αφορά τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και την οικονομική διακυβέρνηση. Ζητώ συγγνώμη λοιπόν γι' αυτό. Δεν είναι ότι δεν σας θέλαμε εδώ. Ούτε ότι έχουμε εμεί πρόβλημα απόδοση, αλλά είχαμε υπερβολικό φόρτο εργασία. Ζητώ συγγνώμη λοιπόν που κάποιε φορέ χρειάστηκε να συμπτύξουμε το χρόνο που είχαμε διαθέσιμο για εσά. Μα έχετε στείλει πολλά έγγραφα σε μένα, τα οποία έχω προωθήσει. στην Επιτροπή και στην Ομάδα Εργασίας Περιενταγωνισμού. Δεν τα έχετε κάνει όλα τέλεια, πρέπει να το επιθυμίζουμε, ε, που και που. Αλλά έτσι φαίνεται να γίνεται σε όλου του τομεί με του οποίου ασχολείται η Κομισιόν. Αλλά πιστεύω ότι έχουμε καθιερώσει εδώ μια καλή πρακτική και ελπίζουμε ότι θα συνεχίσει. Ένα από τα πράγματα που χρειαζόμαστε είναι ένα έγκαιρο πρόγραμμα εργασιών τη Κομισιόν, ειδικά στον τομέα του ανταγωνισμού, έτσι ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπορεί να προγραμματίσει τι δράσει του περί πολιτική ανταγωνισμού. Επίσης θα θέλαμε να καλείται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμμετέχει σε συνεδριάσει με εθνικούς εμπειρογνώμονες για την εκπόνηση νομοθετικών και μη νομοθετικών μέσων. Καλό θα ήταν αυτό να γίνεται τακτικά και όχι κατά εξαίρεση. Όχι κάτι που πρέπει να ζητάμε κάθε φορά. Φυσικά έχει σημειωθεί τεράστια πρόοδος όσον αφορά την οδηγία ε, για αξιώσεις αποζημίωσης ε, στην νομοθεσία ανταγωνισμού και ελπίζουμε ότι θα ολοκληρωθεί ο τριμερής διάλογος. Ελπίζουμε να κλείσουμε το θέμα σήμερα το απόγευμα. Το έχουμε ζητήσει εδώ και πολύ καιρό και από την τελευταία θητεία και είχαμε πει ότι επειδή πρόκειται για ένα θέμα ε, για το οποίο υπάρχουν πολλές διαφορετικές αποφάσεις. Θέλαμε να αποφασιστεί με απόφαση και ευχαριστούμε που τηρήσατε την υπόσχεσή σας προς το Κοινοβούλιο να πράξετε έτσι. Ελπίζουμε λοιπόν ότι σήμερα το απόγευμα θα καταφέρουμε να κλείσουμε το θέμα ικανοποιητικά. Πιστεύω ότι αυτό θα αποτελέσει και ένα εξαιρετικό προηγούμενο Οπότε όταν τελικά προβούμε σε αλλαγή της συνθήκης να συμμετέχει περισσότερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις δημοκρατικές διαδικασίες για θέματα ανταγωνισμού. Αυτό θα γίνει μετά από το λήξη της δικής, της δικής σας Θα απαιτούσε βέβαια αυτό μια γρήγορη αλλαγή της συνθήκης την οποία δεν αναμένουμε. Θα επέλυε βέβαια κάποια προβλήματα. Να επισημάνω ότι έχουμε επιτύχει. Συνεργαστήκαμε με τις υπηρεσίες μας και οι υπηρεσίες, με τις υπηρεσίες σας και οι υπηρεσίες σας συνεργαστήκαν εξαιρετικά με τη Γενική Διευθυνσία Μάρκτ για το σχέδιο κανονισμού των interchange fees, το οποίο επίση αποφασίστηκε με συναπόφαση, πολύ θετική εξέλιξη. Πολλά γίνονται για τις κρατικέ ενισχύσει, Οι προσωρινοί κανόνες κρατικών ενισχύσεων υιοθετήθηκαν από την Κομισιόν στο πλαίσιο της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Ε, είναι οι προμαζόμενες ανακοινώσεις ε, κρίσης. Και είχαμε και τη διαδικασία συγχρονισμού των κρατικών ενισχύσεων. Όσον αφορά την ανακοινώσει για την κρίση, οι κρατικές ενισχύσεις προς τις τράπεζες, η διάρκεια τους και το εξαιρετικό πλαίσιο που τις επέτρεψαν ήταν ένα ε, διαρκώς συζητούμενο θέμα σε διάφορες εκθέσεις της Κομισιόν. Και εμεί αναγνωρίζουμε ότι οι προσωρινοί κανόνε που υιοθέτησε η Κομισιόν να βοήθησαν τη σταθεροποίηση του οικονομικού συστήματο και βοήθησαν ε, στην αποκλιμάκωση τη κρίση ω εργαλείο. Ωστόσο, εκφράστηκαν ανησυχίε για τι συνέπειε που θα μπορούσαν να προκύψουν και για τα κρατικά χρέη. Αλλά αυτό δεν ενταστεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σα. Όσον αφορά τον εξυγχρονισμό των κρατικών ενισχύσεων, επισημάνομαι ότι υπάρχει ανάγκη για λιγότερε και πιο εξυγχρονισμένε, πιο αποτελεσματικέ διαδικασίε. Εδώ βασιστήκαμε στο άρθρο 109 τη Συνθήκη για του δύο κανονισμού του Συμβουλίου που περιλαμβάνουν αυτόν τον εξυγχρονισμό και του κανονισμού ε, εφαρμογή. Εμείς ε, συμβάλαμε ε, επί της ουσίας, αλλά η έλλειψη απόφαση αυτού του τομεί δεν μας ικανοποιεί καθόλου. Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω τον πρόσφατο ρόλο μας στην Διεθνή Συμφωνία με την Ελβετία για την εφαρμογή του ανταγωνισμού, των κανόνων του ανταγωνισμού ε, για τον οποίο συνένεσε το Κοινοβούλιο, παρότι τώρα είναι αβέβαιο κατά πώ θα μπορέσει να διατηρηθεί μετά από το πρόσφατο δημοψήφισμα στην Ελβετία. Αυτός είναι ένας τομέας ε, στον οποίο η Επιτροπή ΕΚΟΝ υποστήριξε πάντα στεναρά τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και στο ευρωπαϊκό δίκτυο ανταγωνισμού και σε διεθνές επίπεδο διότι σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον τα καρτέλ ε, λειτουργούν διασυνοριακά και οι συγχωνεύσεις συχνά εντάσσονται σε πολλές ε, δικαιοδοσίες Ελπίζω λοιπόν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συμμετάσχει περισσότερο στο μέλλον στις διαπραγματεύσεις, στην εκπόνηση κανονισμών για μελλοντικές συμφωνίες ανταγωνισμού. Συνολικά πιστεύω είναι πολύ θετικό που μπορούμε να πούμε ότι συνεργαστήκαμε καλά κατά τη διάρκεια της θητείας σας. Ε, ξέρω ότι δεν φεύγετε ακόμα, αλλά θα διακόψει το Κοινοβούλιο για τις εκλογές, οπότε δεν θα έχετε την ευκαιρία να ξαναρθεί σε αυτή την Επιτροπή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πιστεύω ότι δίνουμε 8 στα 10 στην έκθεσή σας ε, τέλους θητείας. Και με αυτά έχετε τον λόγο. Ε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ Σάρων για τα καλά σου λόγια. Μετά από πάνω από τέσσερα χρόνια που ήρθα για πρώτη φορά στην Επιτροπή σας και μίλησα στα μέλη της. Ελπίζω ότι στο τέλος της θητείας και η θητεία μου θα διαρκέσει λίγο παραπάνω από τη δική σας. Ελπίζω να ανέβω από το 8 στο 9,5. Δεν έχω ολοκληρώσει ακόμα τη δουλειά μου. Το κοινοβούλιο. Ε, άλλωστε θα είναι εδώ μέχρι την τελευταία μέρα της θητείας μου που ελπίζω ότι θα είναι η 31η Οκτωβρίου. ο ορισμός των νέων ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, των επιτρόπων, ε, των ε, υψηλών αντιπροσώπων κλπ. θα πραγματοποιηθεί εκείνη, θα έχει ολοκληρωθεί εκείνη τη μέρα και έτσι θα μπορέσω να παραδώσω το χαρτοφυλάκιό μου στον διάδοχό μου. Πάντως ήταν εξαιρετική η ευκαιρία να συνεργαστώ με την Επιτροπή σας ε, και χαίρομαι για τον τρόπο που πραγματοποιήθηκε λαμβάνοντας υπόψη τους ε, περιορισμούς ε, της συνθήκης. Το Κοινοβούλιο πρέπει να συμμετέχει πλήρως σε όλες τις αποφάσεις νομοθετικής φύσης. Η συνεργασία μας ήταν ανοιχτή, ειλικρινής και για μένα ήταν πολύ χρήσιμη η συνεισφορά σας και θετική. Να συνοψίσω πού βρισκόμαστε τώρα στο τέλος της θητείας σας. Κατά τη διάρκεια αυτής της τελευταίας συνεδρίασης, τι έχω πάνω στο γραφείο μου για τους επόμενους μήνες. Αναφέρατε την οδηγία για τις ιδιωτικές αποζημιώσεις. Ελπίζουμε η αποψινή, ο αποψινός τριμερής διάλογος να είναι επιτυχής και να υιοθετηθεί η οδηγία αυτή πριν τις ευρωεκλογές. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα προόδου για πλήρη επιβολή του νόμου περί ανταγωνιστικής πολιτικής και από την πλευρά του δημοσίου αλλά και από την πλευρά του ιδιωτικού τομέα που χρειάζεται το νομοθέτημα αυτό για να έχει την δυνατότητα αποζημίωσης σε σοβαρές περιπτώσεις παραβίασης ε, του δικαίου περί ανταγωνισμού. Θέλουμε να έχουμε συνθήκες ίσου ανταγωνισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε αυτό το νομοθέτημα. Ελπίζουμε λοιπόν ότι θα υιοθετηθεί με την ψήφο σας στην Ολομέλεια τον Απρίλιο. Περνάμε δύσκολους καιρούς από οικονομικής πλευράς και αυτό δημιουργεί κάποιες απειλές για την εσωτερική αγορά μας. Η ενιαία αγορά δεν έχει επιτευχθεί στο σύνολό της. Ε, αντιμετωπίζουμε σημαντικές προκλήσεις στον τομέα τηλεπικοινωνιών, στην ψηφιακή οικονομία, στον τομέα ενεργείας, στις υπηρεσίες κλπ. κλπ. Η πολιτική ανταγωνισμού και η ενιαία αγορά αποτελούν ε, δύο στοιχεία του ιδίου στόχου να ολοκληρωθούν οι οικονομίες μας, ε, να περάσουμε στην, ευρωπαϊκή στην οικονομική ολοκλήρωση και να το κάνουμε αυτό προς όφελος των πολιτών μας, των επιχειρήσεών μας, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, Και αυτό συνάδει με το ε, ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο. Θέλουμε λοιπόν ε, η οικονομική ανάπτυξη για τους πολίτες μας και γι' αυτό ακριβώς έχω πιέσει για την ε, επιβολή του δικαίου περιανταγωνισμού. Καταρχάς λοιπόν έχουμε τον χρηματοοικονομικό τομέα. Σημαντική δραστηριότητά μας ε, ήταν η αποκατάσταση του ε, χρηματοπιστωτικού τομέα λόγω της κρίσης και έχουμε επικαιροποιήσει το πλαίσιο κρατικών ε, επιχορηγήσεων που υιοθετήθηκε στην αρχή της κρίσης. Θέλουμε λοιπόν να αποκαταστήσουμε τον τομέα, να αποκαταστήσουμε τις συνθήκες ε, ίσου ανταγωνισμού, να ελαχιστοποιήσουμε το ποσοστό των χρημάτων των φορολογούμενων που θα χρειάζεται για την ε, αποκατάσταση του χρηματοοικονομικού τομέα. Η τελευταία αναθεώρηση των σχετικών κανόνων πραγματοποιήθηκε πέρυσι το καλοκαίρι και εφαρμόζουμε τους κανόνες αυτούς ε, με σχετικά καλά αποτελέσματα. Πολλές τράπεζες ε, έχουν ε, αποπληρώσει ή αποπληρώνουν τα χρήματα που έλαβαν ε, στην αρχή της κρίσης. Σε άλλες περιπτώσεις οι τράπεζες αυτές δεν υπάρχουν πια διότι δεν μπορούσαν να επιβιώσουν στην αγορά ούτε με τις κρατικές επιχορηγήσεις που έλαβαν από τα κράτη-μέλη. Πάνω από 20 περιπτώσεις εκαθαρίσεων τραπεζών είδαμε τα τελευταία χρόνια συνεχίζουμε να εργοζόμαστε σε κάποιους ε, τομείς πάνω στα τραπεζικά συστήματα των προβληματικών χωρών, ε, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Κύπρο, την Πορτογαλία, την Ισπανία. Εφαρμόζουμε αποφάσεις που υιοθετήθηκαν χρησιμοποιώντας όχι μόνο δημόσιο χρήμα, αλλά και ε, πόρους που περνάνε μέσα από τα προγράμματα οικονομικής υποστήριξης των χωρών αυτών. Ε, και είμαστε διατεθειμένοι να ενεργήσουμε σε περίπτωση που είναι αυτό απαραίτητο μετά από τα stress test που πραγματοποιούνται αυτή τη στιγμή. Έχουν λοιπόν υιοθετηθεί οι κανόνες Και δεν βρισκόμαστε πια στην αρχή, στην χειρότερη φάση της κρίσης, ε, αλλά απαιτείται ακόμα η ύπαρξη μέσων δημόσιας υποστήριξης για τις τράπεζές μας, εφόσον οι μέτοχοι των τραπεζών αυτών δεν μπορούν να συμβάλλουν με συστήματα διάσωσης που, που εφαρμόζονται τώρα, ε, χάρη μάλιστα και στην δική σας υποστήριξη. Ανησυχούμε πάντως πάντα για τον χρηματοοικονομικό τομέα και όπως ξέρετε κάνουμε κάποιες σημαντικές έρευνες και όσον αφορά την πτυχή του antitrust. Υπήρξαν κάποιες ε, τράπεζες ε, οι οποίες ε, πρωτοστάτησαν στη χειραγώγηση του δίκτυου LIBOR και Συνεχίζουμε να ερευνούμε την ε, περίπτωση αυτού του καρτέλ, ε, όπως και την ε, χειραγώγηση άλλων δικτών, όπως την περίπτωση με τις ελβετικές τράπεζες και τα παράγωγα. Εξετάζουμε επίσης το θέμα των δικτών αναφοράς των ε, πρώτων υλών, ιδιαίτερα στον ε, τομέα της ενέργειας. Όσον αφορά τα καρτέλ, που είναι ο άλλος, ο άλλος τομέας που θέλω να αναφέρω, είναι οι έρευνες ε, για τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων. Έχουμε υιοθετήσει δύο αποφάσεις μέχρι τώρα που έχουν να κάνουν με το αφρολέξ που χρησιμοποιείται για, τη, για τα καθίσματα αυτοκινήτων και τους ε, ημάντες. Πραγματοποιούνται και άλλες έρευνες ε, και θα αποτελέσουν ε, μέρος του μέρος των εργασιών του διαδόχου μου. Ο τομέας των αυτοκινήτων βρίσκεται στον πυρήνα του βιομηχανικού μας τομέα. Στον τομέα της ενέργειας έχουμε πολλές ε, δραστηριότητες. Έχουμε την ε, υπόθεση Gazprom ε, και τις σχετικές αποφάσεις που ελήφθησαν πριν κάποιες εβδομάδες. Εξετάζουμε και άλλες περιπτώσεις επιθανής κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης σε κάποια κράτη-μέλη, για παράδειγμα στην Βουλγαρία. και βρισκόμαστε στις τελευταίες εβδομάδες ε, μιας ε, πολύ σημαντικής εργασίας να ε, αποφασίσουμε τις κατευθυντές γραμμές για τα κράτη στον τομέα της ενέργειας. Θέλουμε να προωθήσουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να πετύχουμε τους ενεργειακούς και περιβαλλοντικούς μας στόχους με τρόπο συνεπή με τους κανόνες κρατικών επιχορηγήσεων και λαμβάνοντας υπόψη τις συνέπειες της στρατηγικής αυτής ε, και την χρηματοδότηση. Θέλουμε να δούμε τις συνέπειες σε, βασικές, σε βασικούς τομείς της βιομηχανίας μας ε, και θέλουμε τα χρήματα που χρησιμοποιούνται για ε, τον ενεργειακό τομέα να χρησιμοποιούνται σωστά και θέλουμε από την άλλη να αποφασίσουμε ε, ποια στοιχεία είναι συμβατά και ποια όχι με την στρατηγική αυτή. Θέλουμε δηλαδή να εξετάσουμε τις συνέπειες στους τομείς κλειδιά ε, των βιομηχανιών μας. Εξετάζουμε τον τομέα τηλεπικοινωνιών. Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο σημαντικές περιπτώσεις συγχωνεύσεων. Μία στην Ιρλανδία και μία στη Γερμανία σε έναν τομέα που χρειάζεται υποστήριξη επειδή Ζητάμε τεράστιες επενδύσεις για να βελτιωθούν τα δίκτυα μας, να βελτιωθούν οι υπηρεσίες τους απέναντι σε άλλους παράγοντες στην αγορά αυτή που αναπτύσσεται πολύ γρήγορα. Έχουμε τους λεγόμενους over-the-top players που είναι οι σημαντικοί παράγοντες. Θέλουμε όμως ε, μία στρατηγική ε, επενδύσεων στον τομέα αυτών, ε, κάτι που δεν μπορεί να γίνει όμως με βάση τους περιορισμούς στον ανταγωνισμό. Οι δύο αυτές συγχωνεύσεις θα περάσουν και στο γραφείο του Επιτρόπου Ανταγωνισμού τις επόμενες εβδομάδες ή τους επόμενους μήνες. Έχουμε συζητήσει λοιπόν επανειλημμένα το θέμα αυτό και με μέλη της Επιτροπής σας καθώς και με άλλους ευρωβουλευτές. Πρόσφατα υιοθετήσαμε ε, σημαντικές κατευθυντήρες γραμμές για τον αεροπορικό τομέα όσον αφορά τον ανταγωνισμό και τις επιχορηγήσεις και τις τελευταίες εβδομάδες ε, εργαζόμαστε πάνω σε κατευθυντήριες γραμμές ε, για την ε, καινοτομία. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Δεν ε, θα αναπτυχθώ περαιτέρω πάνω στη σημασία του θέματος αυτού. Επικεντρωνόμαστε πάντως στην χρήση των δημοσίων πόρων για τις έρευνες και την Και επίσης υπάρχει η άλλη σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία που συζητιέται στο Κοινοβούλιο με τη δική μας συμβολή, με του Μισελ Μπαρνιέ για την ακρίβεια. Μιλάμε για την νομοθετική μεταρρύθμιση του συστήματος πληρωμών και της σχετικής οδηγίας. Κάτι που συμπεριλαμβάνει ε, το θέμα των ε, τελών. Multilateral Interchange. Έχουμε και την ε, έκθεση Σαλβαμέ, τη συμβολή λοιπόν της Επιτροπής σας Πιστεύω ότι θα έχουμε επιτυχία στο θέμα αυτό και είναι ένα θέμα το οποίο συνάδει με τις ε, έρευνες ε, που κάνουμε σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Ε, εξετάζουμε το θέμα της Visa και της Mastercard. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο του συστήματος πληρωμών μας. Αυτές λοιπόν ήταν οι εισαγωγικέ μου παρατηρήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια, για τη φιλοξενία σας, για τη συνεργασία σας και σας εύχομαι καλή επιτυχία στις επόμενες εκλογές. Εύχομαι στους ε, υποψήφιους, ιδιαίτερα σε αυτούς που ανήκουν στο δικό μου κόμμα και σας ευχαριστώ πολύ. Uh, Ευχαριστούμε. Εγώ είμαι δύσκολη στους βαθμούς μου, κανένας δεν παίρνει παραπάνω από 8 στα 10. Θα δώσω το λόγο καταρχήν στον Παύλο Σάλβακ, μέρος του ΑΛΚ. Ε, ό,τι εμένα δεν μου ευχηθήκατε και πολύ τύχη σε αυτές τις εκλογές, εγώ έχοντας ακούσει την ε, ομιλία σας ε, δεν θα ήθελα να προσθέσω ε, βαθμούς ε, σε αυτούς που σας έδωσε η Πρόεδρος, αλλά ε, έχω παρακολουθήσει πιο πολύ μέσω του τύπου ορισμένα πράγματα, για, για παράδειγμα για την Google. Έχω την εντύπωση ότι πετύχατε περισσότερες παραχωρήσεις εσείς από ότι άλλες ρυθμιστικές αρχές. Η ερώτηση είναι εξή. Αν η περίπτωση αυτή είχε φτάσει στα δικαστήρια, θα είχαμε πετύχει ακόμα περισσότερα. Υπάρχει αυτή η περίπτωση. Δεύτερον, για την MIF, ε, για τα Multilateral, multilateral Interchange Fees, ε, για την οποία είμαι υπεύθυνο. Ε, δεν φαίνεται να υπάρχουν μεγάλες διαφορές ανάμεσα στην Κομισιόν και τη θέση που ψήφισαμε εμείς στο Κοινοβούλιο. Μπορείτε να μου το επιβεβαιώσετε. και ο Επίτροπος Αλμουνία. Πράγματι, δεν πρόκειται να σας στηρίξω στις εκλογές, ε, σας εύχομαι ε, προσωπικό επέδο ότι καλύτερο μπορείτε όμως. Και για σας επίσης κύριε Λάγκε, το ίδιο. Την η περίπτωση Google. πόσο γνωρίζω μόνο μία αρμόδια αρχή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης έκανε έρευνα παρόμοια με τη δική μας. Εμείς ξεκινήσαμε τον Νοέμβριο του 2010. Ε, ήταν η Federal Trade Commission στις ΗΠΑ που ξεκίνησε ε, την ίδια περίπεριοδο, λίγο αργότερα από μας τη δική της έρευνα. Για τα ίδια περίπου προβλήματα η Federal Trade Commission ολοκλήρωσε τις έρευνες της πριν από 15 μήνες, το Δεκέμβριο του 2012. με πολύ μικρές διορθώσεις σε ό,τι αφορά την κατάσταση. Ε, πολύ λίγες μονομερείς παραχωρήσεις εκ μέρους της Google και από τη δική μας οπτική γωνία ήταν δευτερεύουσε αυτές οι παραχωρήσεις. Είναι αλήθεια ότι η κατάσταση Google στις ΗΠΑ ε, είναι, η θέση της είναι πολύ ισχυρή στην αγορά. Όχι όμως τόσο ισχυρή όσο στην Ευρώπη. Στην ε, βορειοαμερικανική αγορά ε, η μηχανή ε, αναζήτηση στην Google έχει ένα μερίδιο 70-75% της αγοράς. Ε, υπάρχουν τουλάχιστον δύο ανταγωνιστές οι οποίοι έχουν ένα σημαντικό μερίδιο της ε, αγοράς. Στην Ευρώπη, ή από την άλλη μεριά, η Google δεσπόζει με ένα ποσοστό πάνω από 90%, ε, με μία μόνο νομίζω, εξαίρεση ευρωπαϊκής αγοράς για λόγους που δεν θέλω να σε εξηγήσω αυτή τη στιγμή. Εν πάση περιπτώσει το μερίδιο αγοράς της Google είναι τεράστιο. Όχι επειδή λείπουν οι ανταγωνιστές αλλά επειδή ε, όσοι χρησιμοποιούμε μηχανές αναζήτησης αυτόματα σχεδόν πηγαίνουμε στην Google και πολύ σπάνια συγκρίνουμε με, το, με τα αποτελέσματα άλλων μηχανών αναζήτησης που είναι πολύ προσβάσιμες κατά τα άλλα με ένα πλήκτρο του υπολογιστή μας. Όμως ε, εμείς αυτομάτως πηγαίνουμε στην Google εδώ στην Ευρώπη. Οπότε δεν θέλω να επικρίνω λοιπόν τι έκανε τη Federal Trade Commission, τα πορίσματά της, η κατάσταση είναι διαφορετική ε, ίσως όχι τόσο διαφορετική έτσι ώστε να δικαιολογεί τη διαφορά μεταχείρισης αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα επισέλθω σε αυτό το θέμα. Εμείς συνεχίζουμε με την έρευνά μας, δεν έχει λήξει η έρευνά μας. Βρισκόμαστε σε μια καινούρια φάση, επεξεργαζόμαστε τις επιστολές που θα αποστείλουμε σε καθέναν από τους επίσημους ενάγοντες για να τους εξηγήσουμε γιατί θεωρούμε ότι η τελευταία εκδοχή των προτάσεων της Google που λάβαμε τέλος Ιανουαρίου μπορεί να ε, ρυθμίσει τα σημεία τα οποία θεωρούμε λογικά εύλογα ε, στις, ε, στα αιτήματα των εναγόντων. Θα απαντήσουμε λοιπόν στους ενάγοντες. Δεν μπορώ να αποκλείσω ότι θα μας αναφέρουν επιχείρηματα τα οποία θα μας αλλάξουν τη γνώμη. Αλλά έχουμε συζητήσει πάρα πολύ, το έχουμε σκεφτεί πάρα πολύ. Δεν μπορώ παρόλα αυτά να αποκλείσω οι ενάγοντες να μας πείσουν ότι η κατάσταση ακόμα και έτσι δεν, είναι, ε, δεν έχει επιληθεί. Το τελικό αποτέλεσμα, πόρισμα της έρευνάς μας ε, θα είναι διαθέσιμο πριν λήξει η θητεία της Επιτροπής. Δεν υπάρχει νομικό όριο, χρονικό όριο, αλλά είμαστε έτοιμοι να τελειώσουμε. Ε, ήταν ήδη πολύ μακρόχρονη αυτή η έρευνα, διήρκεσε με μεγάλο χρονικό διάστημα. Νομίζω ότι ε, γίνεται μια συζήτηση η οποία δεν ερμηνεύεται ορθά πάντοτε. Τι εννοώ. Γιατί για αυτήν, όπως και για άλλες όμως περιπτώσεις, χρησιμοποιείται η πολιτική καταπολέμηση της κατάχρησης δεσπόσας θέσης. Γιατί χρησιμοποιείται το άρθρο 9 του κανονισμού που ε, επιτρέπει να αναζητηθούν νομικές ε, δεσμεύσεις μέσω των οποίων να αρθούν τα εμπόδια στον ελεύθερο ανταγωνισμό. Γιατί σε αυτή την περίπτωση και σε άλλες χρησιμοποιούμε αυτή την οδό και όχι την οδό της απλής απαγόρευσης. Για μια σειρά λόγων ε, οι οποίοι αναλύονται σε κάθε έρευνα και οι οποίοι μπορεί να αλλάξουν κατά τη διάρκεια της έρευνας. Αυτή τη στιγμή όμως δεν βλέπω γιατί θα έπρεπε να αλλάξουν για αυτή τη συγκεκριμένη έρευνα της Google. Διότι είναι καλό να έχουμε ένα τελικό αποτέλεσμα νομικά δεσμευτικό που θα επιλύει τα προβλήματα που έχουμε εντοπίσει κατά τη διάρκεια της έρευνας. Σε ορισμένες περιπτώσεις κατά τη διάρκεια της έρευνας έχουμε αλλάξει προσανατολισμό. Τόσο σε έρευνες που ξεκίνησαν μέσω του άρθρου 7, απαγόρευση δηλαδή, και κάποια στιγμή άλλαξαν κατεύθυνση και πέρασαν στο άρθρο 9, με προτάσεις που καταλήγουν σε, σε, νομικούς σε νομικές δεσμεύσεις. Ε, η Upper Samson, για παράδειγμα, ε, την, την οποία θα δούμε σε μερικές ε, ε, εβδομάδες, ε, για καταχρήση σε θέματα βρεστεχνιών. Ε, Ξεκινήσαμε με το άρθρο 7 και καταλήξαμε στο άρθρο 9 και το αντίστροφο όμως. Ξεκινήσαμε σε άλλες έρευνες από το άρθρο 9 και περάσαμε στο άρθρο 7. Επικρατεί μια σύγχυση. Κάποιοι λένε ότι θα πρέπει κάθε φορά να χρησιμοποιούμε το άρθρο 7 στην πολιτική ανταγωνισμό. Όχι, όχι απαραίτητα. Και τα δύο συστήματα εφαρμόζονται ε, ε από το 2004 και μετά. Το θέμα είναι να λύνουμε τα προβλήματα ανταγωνισμού. Αυτό είναι το ζήτημα. Η άποψή μου είναι ότι τα λύνουμε στο μέτρο του δυνατού. Γιατί ε, η πολιτική ανταγωνισμού ε, δεν μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα, ε, δεν είναι ρυθμιστική δραστηριότητα, ούτε νομοθετική δραστηριότητα, είναι μια δράση εκ των υστέρων για να επιλύει προβλήματα τα οποία έχουν εντοπιστεί σε θέματα κατάχρησης δεσπόσας θέσης. Ευχαριστώ. Um, Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σάντσιος Πεσέδο, παρακαλώ. Η θεσμική σχέση της Επιτροπής μας με τον Επίτροπο για θέματα ανταγωνισμού ήταν εξαιρετική, ή της Κομισιόν με το Κοινοβούλιο σε θέματα ανταγωνισμού ήταν εξαιρετική, ε, χαρακτηριστική από διαφάνεια, ε, θεσμική συνεργασία τόσο με τον Επίτροπο όσο και με τους ε, ε, βοηθούς του. Ως πρόεδρος μιας ομάδας εργασίας κάποια στιγμή θέλω να τονίσω ότι αυτή η σχέση ήταν πραγματικά εξαιρετική, άψογη. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι για πρώτη φορά στην πολιτική ανταγωνισμού το Κοινοβούλιο έχει δυνατότητα να λειτουργήσει ως συνεισηγητή σε μια πρωτοβουλία της Κομισιόν. Είναι σημαντικό λοιπόν το γεγονός ότι ο Επίτροπος τίμησε την δέσμευση που είχε αναλάβει κατά τη διάρκεια της ακρόασης του πριν διοριστεί. Ήθελα να κάνω κάποια σχόλια για ορισμένα ζητήματα. Παρόλο που βρισκόμαστε στο τέλος της θητείας μας. Ο Επίτροπος τα τελευταία πέντε χρόνια απέκτησε πολλή εμπειρία. Έτσι κι αλλιώς είχε εμπειρία για οικονομικά θέματα από παλιότερα. Γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να ζητήσω τη γνώμη του. Πρώτον, είναι σημαντικό να διατηρήσουμε τη διαφάνεια. Ε, είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να παρακολουθήσουμε τις κρατικές ενισχύσεις σε ε, χρηματοπιστωτικά ζητήματα είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε το τι συμβαίνει. Και είναι σημαντικό και πάλι η Κομισιόν να συνεχίσει να μας δίνει λεπτομερείς ε, και πλήρες πληροφορίες για όλη την κρίση και τις επιπτώσεις της στους ε, φορολογούμενους και στα δημόσια οικονομικά. Δεύτερον, το θέμα της Google. Υπάρχουν διάφορα ζητήματα σχετικά ασφαλώς αντί για απαγορεύσεις καλύτερα να ε, καταλήγουμε σε νομικές δεσμεύσεις. Όμως το ζήτημα είναι τι θα γίνει με τις ζημίες, τις βλάβες που έχουν προκύψει. Ίσως θα πρέπει να το σκεφτούμε. Όταν ε, όταν ξαναδούμε τον κανονισμό 1 του 2003. Ε, έχουμε ήδη αρκετή εμπειρία, οπότε ίσως στην αναθεώρηση του θα έπρεπε να λάβουμε και το θέμα των αποζημιώσεων τη ε, των, ε, της βλάβης που έχει προκληθεί. θα πρέπει να ξαναδούμε τις σχέσεις μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού πυλώνα, καθώς επίσης και το ότι οι αρχές ανταγωνισμού θα πρέπει να είναι πραγματικά ανεξάρτητες. Αυτό σημαίνει ότι χρειαζόμαστε συγκεκριμένες προδιαγραφές και ο κανόνας λειτουργίας. Και μετά θα πρέπει οι αποφάσεις να έχουν ε, ισοδύναμο αποτέλεσμα με τις κυρώσεις. Ως τώρα δεν έχει επιτευχθεί αυτό. θα ήθελα να μου πείτε τη γνώμη σας. Και σας συγχαίρω και για την εξαιρετική συνεργασία. Ξανά ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και για την, το δικό σας πνεύμα συνεργασίας για κάτι διάρκεια όλων αυτών των τελευταίων ετών. Ήταν χρόνια έντονα με πολλή δουλειά. Όχι εξαιτία των ζητημάτων που άπτονται άμεσα με την ανταγωνιστικότητα, αλλά γενικότερα για τα οικονομικά, χρηματοοικονομικά και χρηματοπιστωτικά ζητήματα. Ε, και ο κύριος Σάντσες Πρεσέδο ε, έχει, εργάστηκε επίσης εξαιρετικά καλά και δεν το λέω επειδή είναι Ισπανός και επειδή είμαστε από το ίδιο κόμμα ε, πραγματικά και η δική σας δουλειά ήταν άψογη Τώρα, σε ό,τι αφορά την διαφάνεια, σε ό,τι αφορά τις κρατικές ενισχύσεις Κρατικές ενισχύσεις προς τον τραπεζικό τομέα. Όπως γνωρίζετε, κάναμε ιδιαίτερη προσπάθεια να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα του scoreboard με έναν τρόπο ευανάγνωστο και χρήσιμο. Ε, τεράστια ποσά των φορολογουμένων διοχετεύτηκαν στον τραπεζικό τομέα. Και προφανώς ε, το τραπεζικό σύστημα βρισκόταν σε κίνδυνο, η κατάσταση βελτιώθηκε, αυτό φαίνεται, και προσπαθήσαμε τα στοιχεία αυτά να τα δώσουμε μέσω της ιστοσελίδας μας, όχι μόνο σας αλλά και σε όλους τους πολίτες. Ένα άλλο θέμα διαφάνειας, το οποίο το περιλαμβάνουμε και στις νέες κατευθυντήριες γραμμές του πακέτου εξυγχρονισμού των κρατικών ισχύσεων, έχει σχέση με τις απαιτήσει, τις οποίες συμπεριλαμβάνουμε σε αυτές τις κατευθύνσεις γραμμές, ε, ε ενημέρωση του κοινού για οποιασδήποτε κρατικές ενισχύσεις δίδονται στον τραπεζικό τομέα. Αυτή τη στιγμή εισάγουμε απαιτήσει διαφάνειας για όλες τις κρατικές ενισχύσεις που χορηγεί κάθε κράτος μέλος. Παρ' όλα αυτά, ορισμένα κρατημέλη έχουν πολλέ ισχυρέ επιφυλάξει προ αυτήν την κατεύθυνση. Πάντω, εμεί κινούμαστε προ αυτήν την κατεύθυνση στις, ε, στο κείμενο που ετοιμάζουμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Google, και όχι μόνο την Google, πώ ε, οι αποφάσει ε, που λαμβάνονται δύναμη του άρθρου 9 θα μπορούν να περιλαμβάνουν και τις αποζημιώσεις για τις βλάβες που έχουν προκληθεί στα θύματα. Θα πρέπει να το σκεφτούμε στο μέλλον. Είναι ε, εύλογο το ερώτημα. Γιατί είτε η απόφαση ληφθεί τη βάση του άρθρου 7, είτε επί τη βάση του άρθρου 9, ε, η, το σκεπτικό είναι ότι έγινε κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης. Αυτή η, αυτή κατάχρηση ε, ρυθμίζεται μέσω της επέμβασης της αρχής ανταγωνισμού, αλλά τι γίνεται με τις αποζημιώσεις. Σωστό, πρέπει να το σκεφτούμε. Και το τελευταίο το οποίο σχολιάσατε, και συμφωνώ μαζί σας είναι πολύ σημαντικό, θα πρέπει να το δούμε στο μέλλον, στην επόμενη θητεία της ε, Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Είναι αλήθεια ότι οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού του δικτύου αρχών ανταγωνισμού από το 2004 και μετά είναι μια πραγματική επιτυχία. Εφαρμόζουμε τους κανόνες της ε, συνθήκης και αυτή η εφαρμογή θα πρέπει να γίνεται με την ίδια αυστηρότητα από όλους. Και στο μέτρο του δυνατού η εφαρμογή αυτή θα πρέπει να γίνεται με συνέπεια, με τον ίδιο τρόπο από όλους. Είτε πρόκειται για αποφάσεις... τη είτε πρόκειται για αποφάσεις... των εθνικών αρχών, αυτέ θα πρέπει να εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο από όλου. Αυτή τη στιγμή οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού δεν έχουν πάντα τους κατάλληλους απαραίτητους ε, επαρκείς πόρους, ούτε την επαρκή ανεξαρτησία πάντοτε. Είναι, ε, έχουμε κάποιες ανησυχίες για ορισμένα κράτη-μέλη. Ε, έχουμε κάποιες πολύ δύσκολες καταστάσεις σε κάποια κράτη-μέλη, προσπαθούμε να τα βοηθήσουμε σε πολλούς τομεί δεν υπάρχει ευρωπαϊκή νομοθεσία σε ό,τι αφορά τις ε, ελάχιστες απαιτήσει από τους ε, εθνικού ρυθμιστικού φορεί. Ε, στην ενέργεια υπάρχει και στι στις ναι, αλλά σε πολλούς άλλους τομεί όχι. Οπότε θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα για το ALDE, όπως φαίνεται αυτή η εκδήλωση είναι ισπανική. Ραμόν Τρεμόσο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Ευχαριστούμε που έρχεστε ξανά εδώ σε αυτό το κοινοβούλιο και θέλω να σας ευχαριστήσω προσωπικά για την εξαιρετική συνεργασία που χαρακτήρισε την τελευταία πενταετία. Έχω δύο ερωτήσει όσον αφορά την υπόθεση αντιτράστη της Google και το τρίτο σύνολο διορθωτικών μέτρων. Η πρώτη αφορά την παρακολούθηση Εμείς ε, ως εκπρόσωποι της Οργάνωσης Πολιτών ε, έχουμε υποχρέωση να παράσχουμε αναφορά στον Monitoring Trustee όσον αφορά τώρα το μηχανισμό η Google θα καλέσει τους τρεις ανταγωνιστές να εμφανίζουν αποτελέσματα αυτά τα δύο στοιχεία θα μεγιστοποιήσουν τα έσοδα που ελπίζει να αποκομίσει το Google. Έτσι λοιπόν οι νικτές του διαγωνισμού θα είναι ίσως αυτοί που θα δημιουργήσουν τα περισσότερα έσοδα για την Google και όχι αυτοί που παρέχουν τις φθηνότερες τιμές για τους καταναλωτές, όχι οι πιο καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όχι τα πιο καινοτόμα προϊόντα. Πώς είναι λοιπόν καλή αυτή η λύση. Τέλος, κατά την απόψή μου, το τρίτο σύνολο διορθωτικό μέτρο είναι καλύτερο για τους ε, καταναλωτές. Δεν το συζητάω. αλλά ίσως οι τιμές είναι υψηλότερες με τις Google Services. Ε, αν είναι να αυξήσει λοιπόν τα έσοδα του Google με έναν μηχανισμό διαγωνισμών μπορεί να αποκτήσει ακόμη πιο δεσπόζουσα ε, θέση. Οπότε η επόμενη επιτροπή να έχει να κάνει περισσότερη δουλειά επί του θέματος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Τρεμόσα. Ε, δεν μπορώ να σχολιάσω συγκεκριμένες πτυχές μιας έρευνας η οποία είναι ακόμα ανοιχτή. Δεν νομίζω θα έπρεπε να συζητούμε τέτοια πράγματα δημοσίως. Τις προάλλες σε μια συνάντηση και κλεισμένο το θυρών με ορισμένα μέλη αυτής και μιας άλλης επιτροπής του Κοινοβουλίου έδωσα κάποιες ε, λεπτομέρειες διότι ήταν πιο ε, απόρριτη και εμπιστευτική εκείνη η συνάντηση. Εδώ δεν πληρώνουν τα ίδια κριτήρια. για τα όσα αναφέρατε, τα ελάχιστα μπορώ να πω είναι το εξής. Ε, ο διαιτητής, ε, ο οποίος θα είναι υπεύθυνο για την ε, σωστή εφαρμογή της απόφασης όταν αυτή λυθεί, στην περίπτωση Google, αυτός ο διαιτητής θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος, θα διοριστεί από την Κομισιόν, θα πρέπει να είναι ένας διαιτητής ο οποίος θα προετοιμάσει και θα αποστείλει στον Επίτροπο Ανταγωνισμού θα προετοιμάζει και θα αποστέλει τακτικές εκθέσεις, μάλλον κάθε τρίμηνο. Εκθέσεις οι οποίες θα βασίζονται στη δική του προσωπική εκτίμηση της εφαρμογής, της υλοποίησης των δεσμεύσεων, καθώς επίσης και θα περιλαμβάνουν και οποιαδήποτε απάντηση σε ενδεχόμενες ερωτήσεις ή προσφυγές εκ μέρους οποιοδήποτε μεταξύ αυτών, αυτών και των καταναλωτών. Οπότε και οι καταναλωτές θα ε, μπορούν να προσφύγουν στο διαιτητή. Ε, και ε, αυτό συμβαίνει και σε άλλες ε, αποφάσεις που λαμβάνουμε βάσει το άρθρο 9. Υπάρχουν τέτοιου είδου διαιτητές, όχι τόσο γνωστοί, ούτε οι υποθέσεις είναι τόσο γνωστές όσο αυτή της Google, αλλά αυτή είναι η κανόνα του παιχνιδιού. Οποιοδήποτε, οποιοδήποτε άτομο ή φορέας έχει κάτι σοβαρό να πει σε σχέση με την μη υλοποίηση ε, ή με κινδύνους μη υλοποίηση απόφαση που έχει ληφθεί επί τη βάση του άρθρου 9 μπορεί να το κάνει. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα και μπορώ να σας πω ότι πραγματικά ο, ο τραστή, ο διαιτητής θα έχει καθήκον να λάβει υπόψη αυτές τις προσφυγές. Ε, πέρσι είχαμε μία μοναδική περίπτωση μη υλοποίηση των δεσμεύσεων απόφαση από τη βάση του άρθρου 9 και η απόφαση ελήφθη πάρα πολύ γρήγορα. πολύ σύντομα μετά την άφηξη των πληροφοριών λάβαμε απόφαση και φρενάραμε ε, την ε, μη εφαρμογή, τη μη υλοποίηση, επιβάλλοντας και πρόστιμο 561 εκατομμυρίων ευρώ. Οπότε ε, βλέπετε ότι ο διαιτητής έχει τη δυνατότητα, έχει τις αρμοδιότητες να επιτηρεί την εφαρμογή. Το σε αφορά τη, τα, την αύξηση των εσόδων μέσω δημοπράτησης. για τις ε, κατακόρυφες αναζητήσεις εξειδικευμένων ε, μηχανών αναζήτησης που ανταγωνίζονται με τις μηχανές αναζήτησης Google. η πληρωμή δεν είναι το ποσό το οποίο προσφέρεται στη δημοπράτηση. Η πληρωμή είναι πληρωμή ανά κλικ, pay per click. Δηλαδή μόνο όταν ο χρήστης πραγματικά κάνει κλικ πάνω στο ε, ε, link το οποίο εμφανίζεται. Ε, όχι δεν πληρώνεται η εμφάνιση, πληρώνεται μόνο το κλικ. Εν πάση περιπτώσει, το επιχείρημα ότι με την παρούσα πρόταση αυξάνονται τα έσοδα της Google δεν με βρίσκει σύμφωνο. Διότι ε, όσο δεν υπάρχουν ανταγωνιστές, ε, η, η Google ε, έχει κέρδη από αυτή την απουσία. ε, αυτά τα χρήματα θα μοιραστούν ανάμεσα στις μηχανές αναζήτησης Google και των ανταγωνιστών. Ανέμενα τη τέλος της ερμηνείας. Τώρα για τους πρασίνους, Μπες Άικοντ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον κύριο Επίτροπο. Θέλω να συζητήσουμε δύο ζητήματα. Το πρώτο αφορά την κρατική ενίσχυση για το με τι ενέργεια και το άλλο αφορά κρατικέ ενισχύσει για ένα αεροδρόμιο στι κατοχώρε από όπου έρχομαι. Για την ενέργεια, στι προτάσει σα πέρυσι δηλώσατε σαφώ ότι η τεχνολογική ουδετερότητα αποτελεί πυρήνα της πρότασης εγώ έχω να πω ότι η τεχνολογική ε, ουδετερότητα όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δοκιμάστηκε στις κατοχώρες από το 2008 μέχρι σήμερα και έτσι αυξήθηκαν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από το 3% σε ένα εντυπωσιακό 4% το οποίο δείχνει σαφώς ότι αυτή η πολιτική τεχνολογικής ιδιωτερότητας δεν λειτουργεί καθόλου και εσεί είπατε ότι αποσκοπεί στο να επιτύχουμε του ευρωπαϊκού στόχου προωθώντα ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια και εγώ ξεκολουθώ να αναρωτιέμαι προ ποια κατεύθυνση κινείστε. Κοιτώντα τώρα τα νέα σχέδια που βρίσκονται σε διπηρεσιακέ διαβουλεύσει που φυσικά κανεί δεν έχει δεκτό από όλου εδώ, υπάρχει πιο μεγαλύτερο περιθώριο για τις μελλοντικέ μακροπρόθεσμες δυνατότητες των νέων τεχνολογιών κάποιες άλλες κατευθύνσεις που θα μπορούσαμε να λάβουμε υπόψη, αλλά θέλω εσείς να μας πείτε τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Για παράδειγμα, αν έχουμε μια, μια μακροπρόθεσμη τεχνολογία που ακριβένει με τα χρόνια, αυτή είναι η πυρηνική ενέργεια. Θα με ενδιαφέρει λοιπόν να ακούσω την άποψή σας για αυτό το σύστημα υποστήριξης του Ηνωμένου Βασιλείου. Θα ήθελα την άποψή σας γι' αυτό. Και τέλος, όσον αφορά τι κρατικέ ενισχύσει για την ενέργεια, πότε θα το προτείνετε. Διότι έξω την ημερομηνία 9 Απριλίου, αλλά αν δείτε τι προέκυψε από τι διαβουλεύσει, είχατε πάνω από χίλιε συμμετοχέ. πιστεύω ότι πρέπει να χρησιμοποιήσετε το χρόνο και να σκεφτείτε έξυπνα για το πώ θα χρησιμοποιήσετε τι ανανεώσιμε αντί να βιαστείτε. Η δεύτερη ερώτηση αφορά ένα αεροδρόμιο στι κάτω χώρε, πολύ κοντά στα γερμανικά σύνορα, πολύ κοντά στο αεροδρόμιο του Μίνστερ Όσταμπρουκ. 100 χιλιόμετρα από εκεί και η Ολλανδική κυβέρνηση παρέχει τεράστιες κρατικές ενισχύσεις ώστε να ε, δραστηριοποιηθεί περισσότερο αυτό το αεροδρόμιο. Ήδη 20 εκατομμύρια και εντός 100 εκατομμυρίων στη γερμανική πλευρά υπάρχει ένα υποεξυπηρετούμενο αεροδρόμιο το οποίο λειτουργεί με ελλείμματα. Και θυμάμαι ότι υπήρχε μια υπόθεση όπου δύο αεροδρόμια ότι δεν μπορεί να δοθεί η κρατική ενίσχυση σε ένα αεροδρόμιο που βρίσκεται 100 χιλιόμετρα, λιγότερο από 100 χιλιόμετρα από ένα άλλο αεροδρόμιο που λειτουργεί ελληματικά. Ήθελα λοιπόν την άποψή σα γι' αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Να αναφερθώ καταρχάς στις περιβαλλοντικές κατευθυντήρες γραμμέ και στην τεχνολογική ουδετερότητα που είναι πολύ καλή αρχή αυτή καθ' αυτή αλλά στην πράξη είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί. Το αναγνωρίζουμε αυτό, δεν έχω εδώ το τελευταίο κειμένο του σχεδίου αλλά όπως είπατε περνάει τώρα διυπηρεσιακή ε, διαβούλευση μετά από μια πολύ ευρεία διαβούλευση και να είστε βέβαιος ότι όλες οι απαντήσεις που θα λάβουμε μέσω που λάβαμε μέσω της ε, δημόσιας διαβούλευσης που ήταν πολύ, πάρα πολλές, εξετάζονται από τις υπηρεσίες μας δεν έχουμε απεριόριστο δυναμικό, αλλά με το περιορισμένο δυναμικό που έχουμε λειτουργεί πάρα πολύ καλά η υπηρεσία μας και είμαι απολύτως ικανοποιημένος με τον τρόπο που έχουν λειτουργήσει οι υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης για, για τον ανταγωνισμό, ιδιαίτερα στο θέμα των κατευθυντηρίων γραμμών που έχουν να κάνουν με την ενέργεια και το περιβάλλον. Πιστεύω πάντως ότι θα διατηρήσουμε την 9η Απριλίου ως ημερομηνία υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών. Θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιουλίου φέτος και πριν τεθούν σε ισχύ θα πρέπει να υιοθετηθούν και να διαδοθούν σε αυτούς που θα πρέπει να τις εφαρμόσουν. Όσον αφορά το θέμα της τεχνολογικής ουδετερότητας, αυτή αποτελεί καλή αρχή, αλλά είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί. Προσπάθησα να καταλήξουμε στο κείμενο που περνάει τώρα από την υπηρεσιακή διαβούλευση να εξετάσουμε τις πιθανές λύσεις και να τις δοκιμάσουμε σε πιλωτικά προγράμματα. Ελπίζουμε έτσι ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στον υψηλότερο δυνατό βαθμό τεχνολογική ουδετερότητα. Ε, σε κάποιε περιπτώσει όμως δεν είναι δυνατόν να υπάρξει κάτι τέτοιο. Αναφερθήκατε στο Ολλανδικό παράδειγμα. Οι κάτω χώρε δεν είναι η μόνη χώρα της Ευρώπης. Υπάρχουν ε, και άλλες εμπειρίες, άλλα στοιχεία, άλλες απόψεις που μας δείχνουν ότι μπορούμε βαθμιαία και ρεαλιστικά να προχωρήσουμε προς μια αρχή η οποία είναι πολύ καλή. Επίσης, ε, πραγματοποιείται έρευνα οι Βρετανικές ε, αρχές εξετάζουν το θέμα αυτό της ε, πυρηνικής μονάδας στο Χίνκλι. Ξεκινήσαμε, ανοίξαμε τον φάκελο τον περασμένο Δεκέμβριο. Οι Βρετανικές αρχές θέλουν να επιταχύνουν τη διαδικασία όσο γίνεται περισσότερο για να ληφθεί η απόφαση, αλλά γνωρίζουν πολύ καλά ότι είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη η περίπτωση αυτή και θα πρέπει να εφαρμόσουμε άμεσα τις διατάξεις της συνθήκης για να αποφασίσουμε με βάση ποια κριτήρια θα κρίνουμε την συμβατότητα ή μη του προγράμματος αυτού ή τις προσαρμογές που θα χρειαστούν στο πρόγραμμα για να θεωρηθεί συμβατό, διότι ούτε στις παλιές ούτε στις ε, νέες κατευθυντές γραμμές δεν συμπεριλαμβάνεται η πυρηνική ενέργεια. Εφαρμόζουμε την συνθήκη, κάτι που αυξάνει τις δυσκολίες στη δουλειά μας, διότι υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία γύρω από την πυρηνική ενέργεια τα οποία δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Εάν μπορέσουμε να υιοθετήσουμε την ε, τελική απόφαση κατά ε, το τέλος της ε, θητείας αυτής της Κομισιόν θα το προτιμούσα. Θα προτιμούσα να μην αφήσω στον διάδοχό μου μια τέτοια έρευνα. Εάν όμως κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν θα συνεχίσουμε τις έρευνες και κατά τη διάρκεια της επόμενης θητείας της Κομισιόν. Όσον αφορά το αεροδρόμιο που αναφέρατε, δεν γνωρίζω την υπόθεση αυτή. Ξέρετε ότι πρόσφατα υιοθετήσαμε τις νέες κατευθυντήρες γραμμές για τα αεροδρόμια και τις αεροπορικές εταιρείες ε, που περιλαμβάνουν σαφή κριτήρια σχετικά με τον τρόπο που κρίνει κανείς ε, το εάν ε, συμμορφώνονται οι επενδύσεις ε, στα αεροδρόμια. Και έτσι εξετάζεται η επιλεξιμότητα των επιχορηγήσεων. Έχουμε κάποιες ε, περιπτώσεις ε, για τις οποίες αναμένονται απαντήσεις με το που θα τεθούν σε ισχύ νέε ε, γραμμές, γραμμέ, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και κατά πόσο ένα αεροδρόμιο μπορεί να αντικαταστήσει άλλα στην περιοχή. Σε μια περιοχή με λογική αυτή να γύρω από το κάθε αεροδρόμιο. Και θα πρέπει να εξετάσουμε όχι μόνο τα άλλα αεροδρόμια, αλλά και τους άλλους τρόπους μεταφοράς, ώστε να διασφαλίζεται η διασύνδεση για τους επιβάτες. Και στην περίπτωση που αναφέρατε, τα δύο αεροδρόμια βρίσκονται πολύ κοντά και το ένα, το παλιό αεροδρόμιο δηλαδή, επιχορηγείται με εθνικούς και ε, ε, ε, πόρους και καθώς και πόρους από τα διευθυντικά ταμεία και επίσης δεν λειτουργεί στο πλήρες δυναμικό του. Και νομίζω ότι η απόσταση 30-35 χιλιόμετρα. Εσείς αναφέρατε μια απόσταση 100 χιλιόμετρων. Ίσως θα κοιτάξω την κατάσταση αυτή, την περίπτωση αυτή. Μάλλον θα είναι στον κατάλογο των περιπτώσεων που αναμένουν απόφαση ή που θα κοινοποιηθούν σύντομα. Μπορώ να σας απαντήσω γραπτός. Ε, ευχαριστώ. Θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο αυστηροί, διότι τελειώς δεν θα προλάβουν όλοι να μιλήσουν. Ο Βέρνερ Λάγγεν. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Επίτροπε. Τέταρτη θητεία μου είναι στην Επιτροπή Οικονομικών. Πρέπει να σας επενέσω. Είσαστε ο πρώτος από το 1994 που λαμβάνει σοβαρά τις διαπραγματεύσεις. Ε, θα ήθελα λοιπόν να σας επενέσω γι' αυτό. Ο Κάλ Φανλιμίαρτ ήταν ε, ε, σοσιαλιστής πραγματιστής, ο Μάριο Μόντι Ιταλός καθηγητής, είναι ελικρούς απλά κοινοποιούσε τις αποφάσεις ε, των ε, υπαλλήλων της ε, χωρίς να διαπραγματεύεται. Είσαστε λοιπόν ο πρώτος που το κάνει αυτό. Θα ήθελα λοιπόν να σας επενέσω που παίρνετε στα σοβαρά τον διάλογο με το Κοινοβούλιο. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Η μία έχει να κάνει με την οδηγία επιχορηγήσεων για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. και υπάρχει ε, γερμανικός νόμος για τις ε, ε, βιώσιμες πηγές ενέργειας που αναφέρεται επίσης στις επιχορηγήσεις και είπατε ότι υποβάλλατε νέα πρόταση όσον αφορά την εσωτερική αγορά, λαμβάνοντα υπόψη δηλαδή τον ανταγωνισμό όχι μόνο εκτό Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και εντός. Και αναφέρεται εδώ το ποσοστό του 20% η ε, ε, η ίδια παραγωγή ενέργειας ε, δεν θα πρέπει να απελευθερωθεί τελείως. Θα σας παρακαλούσα να μας πείτε λίγα λόγια για τη διαδικασία αυτή. Το δεύτερο θέμα που θέλω να αναφέρω ήδη αναφέρθηκε. Έχει να κάνει με την οδηγία για τις αερομεταφορές. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις θα μπορέσετε να τις ολοκληρώσετε μέχρι τον Οκτώβριο με βάση τις νέες κατευθυντήρες γραμμές. Αυτή είναι η δεύτερη ερώτησή μου και η τελευταία ερώτηση μου στο πλαίσιο αυτό αφορά ένα περιφερειακό πρόβλημα. Το κοινό δεν γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα πολιτικής ανταγωνισμού, παρότι αποτελεί θεμελιώδη λίθο στην ε, ευρωπαϊκή κοινότητα. Κάποιο ε, λοιπόν είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κύριο ε, Αλμούνια μας αναγκάζει να ξεπουλήσουμε ε, διότι αλλιώ θα έπρεπε να κλείσουμε την μονάδα, είπε ένα διευθυντή. και πιστεύω ότι μπορούμε να διαδώσουμε καλύτερα την πολιτική ανταγωνισμού στα κράτη-μέλη. Τι μπορεί να κάνει η Κομισιόν για να αποφύγει παρόμοιε περιπτώσει στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λάγκεν για τα γενικά σας λόγια. Φυσικά όπως γνωρίζετε από το 2004, όχι μόνο σε αυτή τη θητεία αλλά και στην προηγούμενη διμερή μας ε, συνεργασία ανέκαθεν υπήρξε καλή. Παρότι όπως συμβαίνει με την υποθέτηση του κ. Θάλμπα και κάποιους άλλους δεν σας υποστηρίζω στις κατευθύνσεις σας αλλά συνεχίζουμε να είμαστε φίλοι. Όπως λέτε η πολιτική ανταγωνισμού δεν είναι πολύ δημοφιλής. Αν σας υποστηρίξω λοιπόν ε, ε, θα δώσω ψήφους στους άλλους. Όσον αφορά την ενέργεια, πέντε είναι τα κυρία σημεία σε αυτές τις γραμμές για την ενέργεια. Πρώτον, δημόσια υποστήριξη στις ε, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ε, δημοσία στήριξη σύμφωνη με τους κανόνες ε, της ενεργειακής υποδομής, σύμφωνη με μέτρα ενεργειακής απόδοσης, πώς να έχουμε συμβατότητα με την υποστήριξη των μηχανισμών ε, δυναμικότητας και το πέμπτο σημείο, τρόπο ειδική αντιμετώπισης. Πώς αντιμετωπίζουν τον τρόπο ειδική αντιμετώπισης που γίνεται σε ορισμένες χώρες στους ενεργοβόρους χρήστες που δεν μπορούν να καταβάλουν την πλήρη χρέωση που ζητείται από όλους τους άλλους χρήστες ενέργειας ηλεκτρικού ρεύματος διότι ε, αυτές οι βιομηχανίες καταναλώνουν υπερβολικά μεγάλες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας. Το έχουμε συζητήσει αυτό με τους διαφορούς τομείς. Θα το συζητήσουμε σήμερα. Έχω δύο συναντήσεις μετά από αυτή την ε, συνάντηση με τομείς που επηρεάζονται άμεσα από αυτή τη διάταξη των κατευθυντήρων γραμμών. Συζητάμε και διαπραγματευόμαστε επίση και με τα κρατη και η Γερμανία είναι ένα από αυτά. Και ξέρω ότι παρότι δυστυχώς ε, δεν καταλαβαίνω τι γράφει ο γερμανικός τύπος κάθε πρωί, γνωρίζω ότι καθημερινά το όνομά μου δεν μπορεί να μεταφραστεί στα γερμανικά, οπότε βλέπω η Αλμούνια και ξέρω ότι μιλάνε για μένα. Προσπαθούμε να καταρτήσουμε έναν κατάλογο τομέων που μπορούν να, να έχουν μερική εξαίρεση των υπερχρέωσεων. Και οι φόροι μπορούν να εφαρμοστούν, το φορολογικό καθεστώ μπορεί να εφαρμοστεί με τον ίδιο τρόπο. Αυτοί οι τομεί θα πρέπει να επιλεγούν βάσει τη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματο. Τι κόστο δηλαδή έχει το ηλεκτρικό ρεύμα και την ποσότητα των συναλλαγών. Διότι για να καταλάβουμε τις συνέπειες για την εσωτερική αγορά και για να αιτιολογήσουμε αυτή την εξαίρεση πρέπει να καταλάβουμε την εξωτερική έκθεση αυτών των τομέων και τους κινδύνους εξαγωγής ε, ε, ανθρακούχων εκπομπών σε άλλα κράτη-μέλη κτλ. Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματο και ποσότητα ε, συναλλαγών. Αυτό είναι το πρώτο, η πρώτη σκέψη και μας οδηγεί σε μια μεγάλη λίστα τομέων. Το δεύτερο στοιχείο είναι πόσο μεγάλη μπορεί να είναι η εξαίρεση. Ω Γενική Αρχή στις κατευθυντήρες γραμμές ε, λέγεται ότι η εξαίρεση θα υπερβαίνει κατά τη την χοντρική ε, προστιθέμενη αξία. Αλλά σε ορισμένους τομείς υψηλής κατανάλωσης θα χρειαστεί ειδική αντιμετώπιση. Αυτή τη στιγμή εμείς ε, ζυγίζουμε τα πράγματα για να δούμε σε ποιο βαθμό θα παρέχουμε τέτοια ειδική μεταχείριση και τι είδου πιο ευνοϊκή μεταχείριση θα μπορούσαμε να παράσχουμε σε αυτέ τι ε, επιχειρήσει υψηλή κατανάλωση ενέργεια ή με μεγάλη έκθεση εμπορική. Δεν έχουμε φτάσει σε τελικά αποτελέσματα Ακόμη και αν ε, μόλις 9 Απριλίου θα λάβουμε την απόφαση, μέχρι τελευταία στιγμή θα πρέπει να ζυγίζουμε τις διάφορες πληροφορίες που λαμβάνουμε, ώστε να εξισορροπήσουμε και να επιτύχουμε επαρκές επίπεδο αποδεκτό εξαιρέσεων. Πάντας υπόψη όλες τις βιομηχανίες και όλα τα κράτη-μέλη διότι οι υπόλοιπε βιομηχανίε θα πληρώσουν όσα δεν πληρώσουν ε, οι εξαιρούμενε βιομηχανίε. Και πρέπει να σκεφτόμαστε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, χωρί να λαμβάνουμε όπω μόνο ένα κράτο μέλο. Αλλά είμαι βέβαιο ότι θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε έναν ε, καλό συμβιβασμό. Όπω είπατε, μου αρέσουν οι διαπραγματεύσει. Ε, και μου αρέσει να διαπραγματεύομαι ό,τι είναι διαπραγματεύσιμο, όχι ότι δεν είναι. Α δούμε λοιπόν πώ θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε μια καλή συμφωνία. Τώρα για τι αεροπορικέ εταιρείε έχουμε διάφορες εκκρεμώσεις υποθέσεις. Την ημέρα που υιοθετήσαμε τις κατευθυντήριες γραμμές, υιοθετήσαμε και κάποιες ε, αποφάσεις βασισμένες αυτές. Τώρα τις επόμενες μέρες θα εγκρίνουμε μια δεύτερη, μια δεύτερη ομάδα αποφάσεων. Θα προσπαθήσω να το επιταχύνω, αλλά δεν μπορώ να προβλέψω αν 31 Οκτωβρίου στα μεσάνυχτα θα υπάρχουν εκκρεμούς υποθέσεις και πώς θα είναι. Θα εξαρτηθεί με τις ανανόσιμες ε, δεν θα συζητήσω με το άτομο για την ε, νομοθεσία στη Γερμανία. Εγώ δεν τη γνωρίζω, την ξέρετε πολύ καλά γιατί την έχουμε συζητήσει πολλές φορές Ποια είναι τα κριτήριά μας όσον αφορά την Green και την έρευνα. όπως σας είπα, την τελευταία φορά που συναντηθήκαμε στο Στρασβούργο, Δεν θα εξετάσω την υλοποίηση τη νομοθεσία περί στη Γερμανία, αλλά όσοι την εφαρμόζουν, αυτοί πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά τι δικέ μα αποφάσει και το δικό μα νομικό πλαίσιο. Καμία συζήτηση λοιπόν ε, υπό αυτού του όρου. θα πρέπει να εφαρμόσει το δικό του νομικό πλαίσιο, το οποίο πρέπει να τηρεί τις διατάξει του δικού μα ε, πλαισίου και αντιστρόφως. Εγώ δεν πρέπει να παρέμβω κατά κανένα τρόπο Τώρα το πώ θα εφαρμοστεί η νομοθεσία στη Γερμανία εναπόκειται στους αρμόδιους στη Γερμανία. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Έχουμε πέντε ε, ομιλητές ε, και 20 λεπτά. Πρέπει να βιαστούμε λοιπόν. Έχω να προτείνω να κάνουμε ένα σύντομο κύκλο ερωτήσεων και απαντήσεων ώστε να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα ώστε να μπορέσουμε να τελειώσουμε εντός της προθεσμίας σε λύσα. Θα μιλήσω αγγλικά για να είμαι πιο γρήγορη. Η ερώτηση μου αφορά τις κρατικές ενισχύσεις και του κανόνες ανταγωνισμού. Συγκρίνοντας το, την εξηγένση των τραπεζών ε, εντός και εκτός του, του τραπεζικού συστήματος, όπως γνωρίζετε είμαι εισηγήτρια για τον ενιαίο μηχανισμό ε, των τραπεζών, ε, θέλω να σχολιάσω δύο πράγματα. Στην ε, EBRD ε, θα έχουμε εργαλεία σταθεροποίησης τα οποία θα χρησιμοποιούνται ε, προκειμένου όταν μια τράπεζα βρίσκεται σε ιδιαίτερες συνθήκες να βοηθηθεί ε, για να περιουστούν οι ζημιές που προκύπτουν. Αυτά τα εργαλεία δεν θα είναι διαθέσιμα μέσα στον ενιαίο μηχανισμό ε, εξυγίανσης, Ούτε η δική μας πρόταση είναι αυτή, ούτε του Συμβουλίου. Επίσης θα υπάρχουν ε, διαφορές στους όρους χρήσης των πόρων. Ε, στο EBRD έχουμε το 8% των συνολικών υποχρεώσεων αλλά και όρους για την είσοδο του Ταμείου εξυγένσης. Όμως, στον ενιαίο μηχανισμό εξυγένσης υπάρχει μόνο ο πρώτος όρος του 8%. Άρα τα συστήματα είναι διαφορετικά. Πώς ε, θα λειτουργήσει αυτό. Ε, όταν δούμε το σύνολο της ενιαίας αγοράς δεν θα έχουμε κάποιο κίνδυνο ε, διαφορετικής μεταχείρισης εντός και εκτός. Δεύτερο, ε, στις για την εξυγένση. Θέλουμε να δώσουμε ρόλο, ισχυρό ρόλο στην Κομισιόν για την εξυγένση. Όμως η Κομισιόν είναι διατεθειμένη να αυτοοργανωθεί έτσι ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει ενδεχόμενες περιπτώσεις κακής χρήσης ε, των ποσών γρήγορα μπορούμε να βασιστούμε στην Κομισιόν ότι θα οργανωθεί με τέτοιο τρόπο ε, έτσι ώστε να μπορεί να συμμετάσχει αποτελεσματικά και γρήγορα χωρίς να σταματήσει ή να τεθεί σε κίνδυνο η διαδικασία. Εξηγένση, σε ευχαριστω Εν συντομία, γιατί ορισμένα πράγματα από αυτά που είπατε είναι πολύ τεχνικά για να τα συστήσουμε εδώ. Όμως είμαστε, ε, και εγώ και οι υπηρεσίες μου είναι στη διάθεσή σας. Ε, η αρχή είναι η εξή. Έχουμε τους κανόνες κρατικών ισχύσεων για το τραπεζικό σύστημα ε, και για την ε, αναδιάρθρωση τραπεζών αλλά και για άλλου τύπου εξηγένση κλπ. Αυτοί οι κανόνες εφαρμόζονται σε επίπεδο των 28 κρατών μελών. Δεν μπορούμε να ε, έχουμε πιο αυστηρή εφαρμογή επειδή μια τράπεζα ανήκει στην Τραπεζική Ένωση και, μια τράπεζα, και άλλη τράπεζα όχι. Θα πρέπει ε, στην εφαρμογή των ε, κρατικών ισχύσεων να είναι οι κανόνες ίδιοι παρόλο ότι υπάρχει διαφορετικό σύστημα για τις τράπεζες της Τραπεζικής Ένωσης και διαφορετικό για αυτές που είναι εκτός Τραπεζικής Ένωσης. Είναι τεχνικά εφικτό. Ε, δεν ξέρω, στην πράξη θα το δούμε. Θεωρητικά είναι εφικτό. Ίσως πρέπει να ρυθμίσουμε κάποιες μικρές δυσκολίες που θα παρουσιαστούν ε, με πιο λεπτομερή τρόπο. Τώρα, το άλλο στοιχείο. Όπως γνωρίζετε εγώ έχω δώσει, έδωσα μάχη όταν προετοιμάζαμε το, την πρότασή μας για τον νέο μηχανισμό εξυγίανσης τόσο μέσα στην Κομισιόν όσο και με το Κοινοβούλιο έτσι ώστε να προστατεύσω την αποκλειστική αρμοδιότητα της Κομισιόν να εφαρμόζει τους κανόνες ε, κρατικών ισχύσεων. Και αν δεν κάνω λάθος τα καταφέραμε. Ε, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ενίου Μηχανισμού ε, τόσο στην Ορομέλεια όσο και το, το Εκτελεστικό Συμβούλιο ε, δεν πρόκειται να λαμβάνει αποφάσεις πριν η Κομισιόν κάνει γνωστή τη γνώμη της. Όπως ακριβώς συμβαίνει και σήμερα, μόνο που πλέον με έναν ολόκληρο μηχανισμό εξυγίανσης που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο ούτε στη ζώνη του ευρώ. Υπάρχει μόνο σε εθνικό επίπεδο σε ορισμένα κράτη-μέλη. Το θέμα της απόφασης για το σχέδιο εξυγένσης που ξεπερνάει τις κρατικές ενισχύσεις, είναι μετά τις κρατικές ενισχύσεις. Η δική μου προσωπική γνώμη είναι εξή. Υποστηρίζω πλήρως τον Μισελ Μπαρνιέ που λέει ότι δεν θα δεχτώ η Κομισιόν να έχει ε, λευκή επιταγή. Η Κομισιόν θα πρέπει να μπορεί να παρεμβαίνει, αλλά για να παρέμβει χρειαζόμαστε λογικές προθεσμίες. Αν οι νομοθέτες θεωρήσουν ότι η, η, ότι η Κομισιόν θα πρέπει να αποφασίσει σε τρεις ώρες, αυτό δεν θα το δεχτούμε. Ε, το θέμα θα παραμείνει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Κομισιόν, αλλά μη μας στριμώξετε, διότι η Κομισιόν δεν θα στριμωχτεί. Δεν θα δεχτεί να στριμωχτεί. Ευχαριστώ, κυρία Μάλετικ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Για να μην καθυστερήσουμε θα μιλήσω κι εγώ στα αγγλικά. Η σπουδαιότητα του ελεύθερου ανταγωνισμού για την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη είναι αναφεσβητητή. Σίγουρα θα πρέπει να διασφαλίσουμε τη σωστή υλοποίηση της πολιτικής ανταγωνισμού σε όλα τα κράτη-μέλη. Ε, μία από τις συστάσεις για τα κράτη-μέλη από την Επιτροπή είναι να στηρίξουν την οικονομική ανάπτυξη με διακανονισμό πρώτης πτώχευσης. Αυτή είναι μια διαδικασία που έχει εισαχθεί τώρα και στη Δημοκρατία της Κροατίας και παρουσιάζει διάφορα πλέον και μειονεκτήματα. Θα ήθελα να μου πείτε την απόψή σας επί του ζητήματος αυτού και πώς το βλέπετε ως εκπρόσωπος πολιτικής ανταγωνισμού. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις ε, της εφαρμογής. Συγγνώμη, εφαρμογή ποιου πράγματος διακανονισμού πρώτης πτώχευσης. Ε, αυτό το θέμα δεν είναι ζήτημα πολιτικής ανταγωνισμού, είναι ζήτημα κανονισμού. Αλλά εάν εμπλέκονται κρατικοί πόροι, η κρατική ενίσχυση θα πρέπει να συμμετέχει σε αυτό. Εγώ και η Επιτροπή δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε μέσα πολιτικής ανταγωνισμού για να συντάσσουμε εθνική νομοθεσία πτώχευση, πρώτη πτώχευση. Τι δεν μπορεί να κάνει η εθνική νομοθεσία, δεν μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που λειτουργούν ε, οι κρατικέ ενισχύσει στο πλαίσιο τη πολιτική ανταγωνισμού. Πρέπει λοιπόν να, επιτυχάνουμε να επιτυγχάνουμε συνοχή χωρί να παρεμποδίζουμε τι ε, αποκλειστικέ αρμοδιότητε Κομισιόν για επιβολή του ανταγωνισμού. Ε, σε πολλά κράτη-μέλη έχουμε καταφέρει να συνάδουν συνεκτικά αυτά τα δύο νομικά πλαίσια. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Δίνω το λόγο στην κυρία Μακάρθη. Well, I too very much want to... Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Επίτροπο και το προσωπικό του για το εξαιρετικό του έργο. Καταφέρετε να δημιουργήσετε καλές συνθήκες ανταγωνισμού και το καταφέρετε με πολύ χιούμορ, με πάντα διάθεση να συζητήσετε και πήγατε μέχρι τα όρια της εμπιστευτικότητας για να μας ενημερώνετε. Το εκτιμάμε ιδιαίτερα και έχετε δημιουργήσει ένα εξαιρετικό ιστορικό, πιστεύω, Ω πρώην πρόεδρο ε, τη Επιτροπή Καταναλωτών, ε, εγώ θεωρώ ότι έχετε κάνει πολλά για του καταναλωτέ. Ε, αναλάβετε πολλέ δράσει και δώσετε πολλέ επιλογέ αποζημίωση. Επειδή αναφέρετε τα benchmark, τα ορόσημα και θεωρώ ότι όλο και δυσκολεύει αυτό το τομέα για μα. Για την υπόθεση Libor Euribor, οι κανόνε antitrust είπατε ότι είναι συμπληρωματικοί, αλλά δεν είναι απλά συμπληρωματικοί. Εγώ θεωρώ ότι η νομοθεσία είναι ένα όργανο αλλαγής συμπεριφορών. Αλλά πολλοί κόσμοι μπορεί να προσπαθεί να, προ... να παρακάμψει τέτοιου κανόνες. Με αυτό που κάνετε εσείς ε, είναι σαφές ότι αλλάζετε τις συμπεριφορές και αυτό είναι πολύ σημαντικό στον οικονομικό κόσμο. Αλλάζετε την ηθική. Θέλω να μου πείτε λοιπόν, σας απασχολούν άλλοι τομείς ε, εμπορίας αγαθών, ε, έχουμε ζητήσει για τη φορέξη, για το πετρέλαιο, για το φυσικό αέριο. Υπάρχουν σοβαρά ζητήματα εκεί. Όλοι αυτοί οι τομεί αυτών των benchmark που είναι σημαντικοί για τη λειτουργία τη πραγματική οικονομία ε, θεωρώ ότι χρειάζεται περισσότερη εξέταση. Θεωρείται ότι οι τιμέ των. Θεωρείται ότι οι οργανισμοί αναφορά τιμών Εμεί θέλουμε πολύ μεγάλο εύρο. Ε, θεωρούμε ότι πρέπει να συμπεριληφθούν τέτοιοι οργανισμοί, press reporting agencies. Και τώρα μια φιλοσοφική ερώτηση. Τι πιστεύετε ότι πρέπει ακόμα να γίνει κατά τη θητεία σα, Δεν θέλω να μα πείτε τα πάντα, γιατί έχετε μεγάλο χαρτοφυλάκιο, αλλά ποιε είναι οι προτεραιότητέ σα πριν ολοκληρώσετε την θητεία σα. Και ελπίζουμε φυσικά ότι θα την ολοκληρώσετε με επιτυχία, όπω σε όλη τη τη διάρκεια. Και θα ήθελα να μου δώσετε και μια εικόνα για το επόμενο κοινοβούλιο. Ποιοι μελλοντικοί τομεί θεωρείτε ότι θα είναι οι σημαντικότεροι, οι τομεί κλειδιά που θα πρέπει να εξετάσουμε για πιθανέ συμπεριφορέ καρτέλ ή ε, συμπεριφορέ που βλάπτουν τον ανταγωνισμό. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πολύ, κυρία Μακάρτη. Σε ευχαριστώ, ακλιν για τα καλά σου λόγια. Όσον αφορά λοιπόν την ε, πολιτική ανταγωνισμού Πρόκειται για ένα πολύ ισχυρό μέσο. Οι συνέπειες είναι άμεσες και μπορούν να είναι τεράστιες. Είναι όμως ε, ένα μέσο που εφαρμόζεται εκ των υστέρων. Δεν είναι πολύ καλό μέσο αν θέλουμε να προβλέψουμε το μέλλον. Αντιμετωπίζει τις παρούσες περιπτώσεις, τις παρούσες παραβάσεις και προσπαθεί έτσι να καταλήξει στις σωστές αποφάσεις. Αλλά δεν είναι εύκολο να προβλέψουμε το μέλλον. Θα προσπαθήσω να απαντήσω όσον αφορά τις ε, τιμές αναφοράς, ε, τα benchmarks. Ε, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε πάνω στο θέμα αυτό. Έχουμε τρεις τράπεζες και έναν διαμεσολαβητή που εξετάζουμε στην περίπτωση Euribor Libor. Έχουμε κάποιες προκατακτικές εργασίες πάνω στο Forex. Έχουμε και μία έρευνα όσον αφορά τις τιμές αναφοράς ε, στα, ε, στο πετρέλαιο και τα παραγωγά του, μπορεί να έχουμε και άλλες περιπτώσεις ε, στο μέλλον. Πάντως, εάν είχαμε περισσότερους ανθρώπινους πόρους, ίσως θα μπορούσαμε, ίσως θα μπορέσουμε στο μέλλον να ξεκινάμε έρευνες δικές μας και θα συνεχιστούν οι εργασίες μας τα επόμενα χρόνια. Ο επόμενος Επίτροπος Ανταγωνισμού θα επικεντρωθεί τουλάχιστον εν μέρη στις περιπτώσεις αυτές. Δεν μπορώ να αποκλείσω όμως να αμφισβητηθούν κάποια άλλα benchmarks στο μέλλον. Και να εξετάσουμε την περίπτωση χειραγώγησης ε, των ε, τιμών αναφοράς. Όσον αφορά τις ε, προτεραιότητες μας. Φυσικά το θέμα αυτό των παραβάσεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα και ξεπερνάει κατά πολύ τις ικανότητες του νομοθέτη και των ρυθμιστικών άρχων. Θυμάμαι ότι συναντήθηκα με εκπροσώπους του χρηματοπιστωτικού τομέα πριν κάποιους μήνες και ανησυχούσαν ανησυχούσαν ειλικρινά λόγω της έλλειψης εμπιστοσύνης ε, των πολιτών, των καταναλωτών ε, απέναντι στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ε, λόγω των όσων μάθαμε κατά τη διάρκεια της κρίσης. Αυτό όμως δεν είναι απλά θέμα νέας ρύθμισης. Χρειάζεται η νέα ρύθμιση και εργάζεστε και εσείς πάνω σε αυτό. Επίσης δεν είναι μόνο θέμα επιβολής ε, του νόμου περί ανταγωνισμού, ε, είναι επίσης ένα θέμα που μας απασχολεί ε, και οι Αμερικανοί και οι αρχές αντιτράστ ασχολούνται με το θέμα αυτό. Αλλά το θέμα εδώ είναι η ιδεοδολογία του χρηματοπιστωτικού τομέα. Πριν την κρίση ήθελαν πάρα πολύ να μας πείσουν να τους επιτρέψουμε την αυτορύθμιση. Ε, θα πρέπει να ρυθμίσουν ε, όμως ε, την δεοντολογία τους και τα ηθικά τους πρότυπα. Αν συνεχίσουμε εμείς να, ανακαλύψουμε ανακαλύπτουμε τέτοιες περιπτώσεις παραβάσεων, ποιος θα έχει εμπιστοσύνη σε κάποια τιμή αναφορά στην πρακτική μιας, ενός οικονομικού τομέα που βασίζεται στην εμπιστοσύνη. Άλλες προτεραιότητές μας είναι η ενέργεια. Δεν μπορώ τώρα σε λίγα λεπτά να εξηγήσω γιατί, αλλά είναι σαφές ότι η ενέργεια είναι τομέας κλειδί. Και θα πρέπει και οι ρυθμιστές σε ευρωπαϊκό επίπεδο και οι αρχές ανταγωνισμού να ασχοληθούν με το θέμα αυτό. Επίσης, οι τηλεπικοινωνίες και ο ψηφιακός τομέας, καθώς και όλες οι δραστηριότητες που συνδέονται με το διαδίκτυο. που δεν ρυθμίζονται ακόμα. Κάποια στιγμή θα ξεκινήσει η ρύθμιση σε διάφορα επίπεδα, σε διάφορους τομείς, αλλά στο μεταξύ σχεδόν το μόνο διαθέσιμο μέσο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να λύσουμε τα προβλήματα, όπως με την Google. Ανέφερα την ε, περίπτωση καταχρήσεων των ε, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, καθότι τελειώνει ο χρόνος θα ακούσουμε τις ε, δύο τελευταίες ερωτήσεις. Ε, ο Πίτερ Σκίνερ και μετά ο κύριος Κλίνης. Ευχαριστώ Επίτροπε. Ευχαριστώ που μας συναντήσατε και τις προάλλες. Η συνάντηση αυτή και, κλεισμένων των θυρών ήταν πολύ χρήσιμη. Βέβαια την επόμενη μέρα διαβάσαμε στις εφημερίδες το περιεχόμενο. Κρίμα. Γι' αυτό πρέπει να σεβόμαστε λίγο ένα τον άλλο. Εν πάση περιπτώσει, η περίπτωση Google εκκρεμεί. Δεν συμφωνώ πλήρως μαζί σας. Και δεν νομίζω ότι πολλοί από εμά σε εκείνη τη συνάντηση θα συμφωνούσαν μαζί σας. Αλλά πάντως είναι σημαντικό που αναλάβατε κάποιες δεσμεύσεις. Η FTC όπως είπατε ε, δεν παρενεύει πολύ, όμως έχει τη δυνατότητα να ξεκινάει έρευνες όποτε το επιθυμεί. Εσείς όμως έχετε ένα buffer 5 ετών. Γιατί δεν μικραίνουμε αυτή την περίοδο. Αν χρειάζεται να τους εξετάσουμε, να τους ερευνήσουμε, πάντοτε, να μπορούμε. Μετά, Σε ό,τι αφορά το Λίβερπουλ για το ε, ferryboat ε, με τα χρήματα τα οποία δόθηκαν από τα διορθωτικά ταμεία. Τα ποσά αυτά δεν είχαν ως σκοπό να χρησιμοποιηθούν ε, σε τομείς ανταγωνιστικούς. Η κυβέρνηση της Βρετανίας ζήτησε τα χρήματα πίσω, η Κομισιόν κατέληξε διαφορετική απόφαση και δεν ζήτησε ανάκτηση των ποσών. Μπορείτε να μου σχολιάσετε αυτό το ζήτημα. Ε, Mr. Clint left, so... Ο κ. Κλίντ έφυγε, οπότε δίνω το λόγο στον Επίτροπο. Ε, ας ομαδοποιήσουμε τις ερωτήσεις. Α, ας απαντήσει τον κύριο Σκίνερ. Σε ένα λεπτό δεν θα πάρω πολύ. Σε ό,τι αφορά την περίπτωση Google. και εμένα με ανησυχεί το γεγονός ότι ε, το περιεχόμενο μιας ε, κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίασης έγινε γνωστό την επόμενη μέρα. Ε, η πενταετής περίοδος για την υλοποίηση των δεσμεύσεων. Αν παραβιαστούν οι δεσμεύσεις, οι συνέπειες είναι άμεσες και είναι αυστηρές. Δεύτερον, αυτές οι δεσμεύσεις, οι πενταετής δεσμεύσεις αφορούν τέσσερα θέματα, όχι την εταιρεία, όχι την εταιρεία στο σύνολό τη. Η έρευνα, η εταιρεία αυτή ερευνάται και για άλλα θέματα. Παρόλο που μας πρότεινε δεσμεύσεις πενταετής. Οπότε δεν αυτή η πενταετής περίοδος δεν μας περιορίζει. Δεν περιορίζει ε, την δυνατότητα που έχουμε να ε, παρακολουθούμε την εταιρεία αυτή. Η πενταετής περίοδος είναι πολύ λογική και συνήθις ε, περίοδος για την ε, υλοποίηση δεσμεύσεων. Θα παρακολουθείτε από τον διαιτητή, ε, από τις αρχές ανταγωνισμού και με πολλούς τρόπους έχουμε τη δυνατότητα ως Κομισιόν να δράσουμε. Σε ό,τι αφορά την περίπτωση του Λίβερπουλ δεν την γνωρίζω καλά, οπότε δεν μπορώ να σας δώσω απάντηση. Στείλτε μου αν θέλετε το, τα στοιχεία αυτής της υπόθεσης και θα σας απαντήσω. Ευχαριστώ. Ο κ. Κλίμπτ. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Θα είμαι σύντομος. Σε παγκόσμιο, σε επίπεδο έχουμε λίγος πολύ παρόμοιους κανόνες ανταγωνισμού με τις ΗΠΑ. Ε, παρόμοιες αυστηρότητας. Τι γίνεται όμως με τις αναδυόμενες αγορές και το δικό τους δίκαιο ανταγωνισμού, Κίνα κλπ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κλίντς για τη συνεργασία που είχαμε καταρχήν για πολλά χρόνια. Ε, έχουμε πολύ καλές σχέσεις με τις αρχές ανταγωνισμού των υπόλοιπων βιομηχανικών χωρών. Εδώ και χρόνια. Αυτές οι σχέσεις είχαν οικοδομηθεί επί τη βάση ε, μνημονίων ε, συνεργασίας, διμερών επαφών και συμφωνιών συνεχούς τακτικού διαλόγου κλπ. Είχαμε πολλές περιπτώσεις που αφορούσαν τρεις-τέσσερις διαφορετικές αρχές ανταγωνισμού διαφορετικών κρατών. Οπότε το έχουμε συνηθίσει. Και έχει βελτιωθεί και η σύγκληση απόψεων τα τελευταία πέντε χρόνια. Σε ό,τι αφορά τις αναδυόμενες χώρες. Και εκεί επισημοποιούμε τη σχέση μας. Πέρσι υπογράψαμε σύμφωνα συνεργασίας με δύο από τις τρεις κινέζικες αρχές. Με την τρίτη είχαμε ήδη συμφωνία. Τώρα καλύπτουμε και τις άλλες δύο. Έχουμε τακτικές επαφές, διάλογο. Υπογράψαμε με τις Ινδικές αρχές. Στο Δελχή εγώ υπέγραψα αυτή τη συμφωνία πριν από μερικούς μήνες. Έχουμε με τη Βραζιλία, έχουμε με τη Ρωσία παρόμοιες συμφωνίες. Και τώρα προτείνω και στην ε, αρχή ανταγωνισμού της Νότιας Αφρικής να ε, συστήσουμε τέτοιου είδους σχέσεις τακτικές. Επιπλέον έχουμε και δύο πλατφόρμες φορά διαλόγου, τον ΩΣΑ, ορισμένες αυτές τις χώρες συμμετέχουν για την ΕΜΕΛ του ΩΣΑ και όλες εκτός των Κινέζικων ε, συμμετέχουν και στο Διεθνές, Δίκαιο Ανταγωνισμού, ε, Διεθνές Δίκτυο Ανταγωνισμού που δημιουργήθηκε πριν από 11 χρόνια. Είναι μια πολύ χρήσιμη πλατφόρμα ανταλλαγής απόψεων, συζήτησης βέλτιστων πρακτικών, σύγκρισης ε, διάφορων διαδικασιών, ε, συζήτησης συγκεκριμένων ζητημάτων. Οπότε αυτές οι αρχές ανταγωνισμού όλο και περισσότερο εντάσσονται στα δίκτυά μας με ένα πολύ δυναμικό τρόπο. Πάντως ε, δεν έχουν φτάσει σε όλες τις περιπτώσεις να κατακτήσουν την πολιτική ανεξαρτησία που είναι απαραίτητη για την καλή εφαρμογή της, ε, του δικαίου ανταγωνισμού. Πολύ συχνά η νομοθεσία περί ανταγωνισμού είναι πολύ παρόμοια με τη δική μας εκεί, αλλά σε μερικές περιπτώσεις η πολιτική τους ανεξαρτησία δεν είναι επαρκής προκειμένου να γίνεται αξιόπιστη εφαρμογή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πίτροπε, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την τελευταία ανταλλαγή απόψεων Ε, σας εύχομαι καλή επιτυχία και ε, στο επαγγελματικό και στο προσωπικό. Ευχαριστώ πολύ. Περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, τη δημόσια ακρόαση με την κυρία Ντανιέλ Νούι, που όπως όλοι γνωρίζετε είναι πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αυτή είναι η πρώτη τακτική δημόσια ακρόαση για τον SSM όπως προβλέπετε στη διοργανική συμφωνία. Μια σειρά ερωτήσεων έχουν σταλεί στην κυρία Νούη πριν από την ακρόαση η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα απάντησε με επιστολή της 17ης Μαρτίου. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα στην κυρία Νούη που παρευρίσκεται σε αυτή τη συνεδρίαση και μόλις είστε έτοιμοι μπορώ να σας δώσω το μικρόφωνο για 10 με 15 λεπτά. Yes. Okay. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου. Είναι η πρώτη μου τακτική δημοσία κρόση στην ΕΚΟΝ σύμφωνα με την διοργανική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Κοινοβουλίου. Δεσμεύομαι να εφαρμόσω το γράμμα και το πνεύμα αυτής της συμφωνίας. Πρέπει οπωσδήποτε να διασφαλίσουμε αποτελεσματική και υπεύθυνη ευρωπαϊκή εποπτεία προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών. Αυτή είναι η τελευταία τακτική δημόσια ακρόση για τον ενιαίο μηχανισμό εξηγένσης ε, για αυτή τη θητεία. Σας ευχαριστώ λοιπόν κύριε Πρόεδρε και αγαπητά μέλη και την Επιτροπή ΕΚΟΝ για τον αποφασιστικό ρόλο που διαδραματίσατε στην υιοθέτηση του κανονισμού SSM και στην νομοθετική διαδικασία προς μια ολοκληρωμένη τραπεζική ένωση. Θα ήθελα να καλύψω τρία σημεία σήμερα Πρώτα απ' όλα όσον αφορά τις ε, προετοιμασίες για τον ε, ενίο μηχανισμό, βρισκόμαστε εντός των προθεσμίων. Οι περισσότεροι κύριοι διευθυντές έχουν διοριστεί και ετοιμαζόμαστε να προσλάβουμε τους 800 επόπτες που χρειαζόμαστε επιπλέον. Η σύνθεση των κοινών εποπτικών ομάδων που αποτελούν το θεμέλιο λίθο του συστήματος με ε, την ευθύνη καθημερινής ε, εποπτείας ε, και καθημερινών δραστηριοτήτων για τις τράπεζες έχει αρχίσει να αποκτά μορφή. Δεν έχει οριστεί πώς οι εθνικοί επόπτες θα εκχωρηθούν σε κάθε μία από αυτές τις κοινέ εποπτικές ομάδες. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχεδιάζει λύσεις πληροφορικής που θα υποστηρίζουν τις εποπτικές διαδικασίες και ιδιαίτερα το έργο αυτών των κοινωνιών ομάδων. Σημαίνεται ικανοποιητική πρόοδο για ισχυρή και ανθεκτική συνδεσιμότητα με τους 7 ε, εθνικούς επόπτες που δεν είναι κεντρικοί τραπεζίτες. Η ΕΚΤ θα δημοσιεύσει μέχρι 4 Μαΐου του 2014 τον κανονισμό μετά από δημόσια διαβούλευση που μόλις ολοκληρώθηκε. Έχουμε ήδη αναπτύξει σε μεγάλο βαθμό το εποπτικό μοντέλο του SSM που ορίζεται στο σχετικό εγχειρίδιο. Το εγχειρίδιο αυτό καλύπτει τις γενικές αρχές, τις διαδικασίες καθώς και τη μεθοδολογία εποπτείας τόσο σημαντικών όσο και λιγότερο σημαντικών τραπεζών. Περιγράφει τη διαδικασία συνεργασίας εντός του SSM και εκτός Το εγχειρίδιο αυτό είναι εσωτερικό έγγραφο του προσωπικού, αλλά εμείς ε, ε, σχεδιάζουμε να εκδώσουμε και μια δημόσια έκδοση. Η προετοιμασία του πέμπτου πλαισίου του ενιαίου μηχανισμού εποπτείας ε, βρίσκεται καθοδόν. Προβλέπεται η πρώτη διαβούλευση στο πρώτο εξάμεινο του 2014, όπου ο κανονισμός για τα τέλη θα τεθεί σε ισχύ τον Νοέμβριο του 2014. Το Εποπτικό Συμβούλιο αυτή τη στιγμή μελετά τους κανόνες διαδικασιών για διοντολογίας Επίσης ο κανονισμός του SSM δεν ζητά ρητά κωδικά δεοντολογίας για τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου. Αναφέρεται σε κάποιους κανόνες ηθικής που θα ισχύουν ιδιαίτερα για αυτούς, όπως αυτοί που αφορούν τη συγκρούση συμφερόντων που απορρέουν από επακολουθή απασχόληση απαιτήσει για τον κώδικα διοντολογία όσον αφορά το προσωπικό και του διοικητέ τη ε, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζας εξεταζονται. επίση θα υποβληθεί πρόταση εν ευθέτω χρόνο στο Εποπτικό Συμβούλιο και στου Οργανισμού λήψη αποφάσεων τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζας μετά από διαβούλευση με του εκπροσώπου του προσωπικού. Πριν την υιοθέτηση, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα ενημερώσει την Επιτροπή ΕΚΟΝ για τα κύρια στοιχεία του προβλεπόμενου κώδικα διοντολογία σύμφωνα με την διοργανική συμφωνία. Επίσης προχωρούν εργασίες για την υλοποίηση τη αρχή διαχωρισμού μεταξύ τη νομισματικής πολιτική και τη εποπτική λειτουργία. Το Εποπτικό Συμβούλιο έχει συζητήσει τη μορφή των διαδικασιών που ολιστικοποιήθηκε πριν από μερικέ μέρες μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αφού εξετάστηκαν πολλές επιλογέ το, το Εποπτικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι θα υποβάλει αρχείο καταγραφή των διαδικασιών τριμηνιαία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό σημαίνει ότι οι διαδικασίε που σχετίζονται με τι συναντήσει από Ιανουάριο μέχρι Μάρτιο θα διαβιβάζονται τέλη Απριλίου, έω τα τέλη Απριλίου. Αλλά το Εποπτικό Συμβούλιο αποφάσισε επίση ότι ο κώδικα εσωτερικών διαδικασιών θα παρέχεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νωρίτερα σε περίπτωση που ζητήσει κάτι τέτοιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είμαι έτοιμο λοιπόν να χρησιμοποιήσω αυτή τη δυνατότητα εάν εσεί θεωρήσετε ότι η τριμηνιαία αυτή διαβίβαση δεν είναι επαρκής. Για να περάσουμε στο δεύτερο σημείο, η ολοκληρωμένη αξιολόγηση προχωρά όλο ταχώς. Να τονίσω ότι η ολοκληρωμένη αξιολόγηση θα είναι αυστηρή. Το κατόφλιο ελέγχου της ποιότητας είναι 8% για το stress test ε, στο βασικό σενάριο. Το κατόφλιο είναι επίσης 8% ε, κεφάλαια κοινομετοχών ε, κατηγορίας 1 ενώ στο αντίξωο σενάριο είναι 5,5%. Αυτά τα κατόφλια είναι υψηλότερα από την προηγούμενη άσκηση. Απαιτούν υψηλότερη ποιότητα κεφαλαίων από το παρελθόν. Επιπλέον, τα stress test θα περιλαμβάνουν κεφαλαϊκέ απαιτήσει που μπορεί να απορρεύσουν από τον έλεγχο ποιότητα του να και του ενεργητικού. Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι πιο απαιτητικό από τι προηγούμενε ασκήσει. Η προετοιμασία της υλοποίησης, της ολοκληρωμένης αξιολόγησης ε, βρίσκονται στον δρόμο τους. Ε, έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των χαρτοφυλακίων που πρέπει να ελεγχθούν. Τώρα βρίσκομαστε στη φάση 2 της άσκησης, την φάση εκτέλεσης. Όσον αφορά τον έλεγχο ποιότητα ε, των περιοριστικών στοιχείων, έχουν εκδοθεί δύο εγχειρίδια στι 11 Μαρτίου. Αυτή η διαφάνεια αυξάνει την αξιοπιστία τη άσκηση, δείχνει την αυστηρότητα και την ολοκληρωμένη τη μορφή να σας δώσω μερικά παραδείγματα για τις 128 τράπεζες που εμπλέκονται στην άσκηση. Συνολικά 760 στην συναλλαγών έχουν επιλεγεί. Ο έλεγχος θα εξετάσει 135.000 αρχεία. Εκτιμάμε ότι χίλια μέλη προσωπικού, εποπτικού προσωπικού ε, και ελεγχού αυτή τη στιγμή έχουν διοριστεί για να υποστηρίξουν τους επόπτες. Ε, πρόκειται για ποσό 3,7 εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή 55% του κεφαλαίου κινδύνου των τραπεζών. Επίσης οι προετοιμασίες ε, για την άσκηση stress τεστ σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση κοντεύουν να ολοκληρωθούν για τη μεθοδολογία και τα σενάρια. Αυτά θα έχουν ολοκληρωθεί και θα δημοσιευτούν τον Απρίλιο του 2014. Για μεγαλύτερη αξιοπιστία της άσκησης χρειαζόμαστε ένα προστατευτικό μηχανισμό σε εθνικό και ως έσκατη λύση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κάνω έκκληση στα κράτη-μέλη να ανανεώσουν την ισχυρή τους δέσμευση και να φροντίσουν να υπάρξουν οι σχετικέ διευθετήσει σε εθνικό επίπεδο συμπεριλαμβανομένων των μηχανισμών εξηγένση και των δημόσιων ανασταλτικών μηχανισμών ώστε να ανταποκρίνεται γρήγορα μόλι εντοπιστεί οποιοδήποτε, ευάλωτο σημείο. Περνάω στο τρίτο και τελευταίο μου σημείο η οδό ε, που θα ακολουθήσει η Τραπεζική Ένωση προς την, την Τραπεζική Ένωση γιατί προς τα εκεί κινούμαστε η πρόοδος ε, υπήρξε γρήγορη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει συμμετάσχει σε αυτή την άσκηση. Πρέπει να διατηρήσουμε αυτή την ταχύτητα. Οι κοινέ προσπάθειες δέσμευσης όλων των απαραίτητων ε, φορέων είναι απαραίτητες ώστε να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση της Τρεπιστικής Ένωσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο τώρα απαιτεί ολοκλήρωση της νομοθετικής διαδικασίας για το SRM σε αυτή τη θητεία ώστε να διασφαλιστεί ότι θα τεθεί σε λειτουργία το σύντομότερο δυνατόν αφού αναλαβεί πλήρε εποπτικέ ευθύνε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Γι' αυτό το σκοπό όλα τα εμπλεκόμενα μέρη θα πρέπει να δείξουν βούληση συμβασμού ώστε να καθιερωθεί ένα πραγματικό ενιαίο μηχανισμό εξυγένση με αποτελεσματική διακυβέρνηση, ενιαίο ταμείο εξυγένση και επαρκή προστατευτικέ διατάξει και διευθετήσει. Για να το πω απλά, όταν καίγεται ένα σπίτι, η πυροσβεστική δεν μπορεί να περιμένει μέχρι να συμφωνήσει το Δημοτικό Συμβούλιο κατά πόσο θα παρέμβει. Όπως λοιπόν μια αποτελεσματική πυροσβεστική χρειάζεται πρόσβαση σε νερό, το SRM χρειάζεται πρόσβαση σε ένα ταμείο επιλύσεις, ε, εξηγήσεις, συγγνώμη. Να τονίσω επίσης ότι η Τραπεζική Ένωση έχει τη δυνατότητα να συμβάλλει σημαντικά την παρολοκλήρωση των οικονομικών χρηματοπιστωτικών αγορών στην Ευρώπη. Σε αυτό το πλαίσιο, ένα κοινό σύστημα εποπτείας και εξυγίανσης αυξάνει τις δυνατότητες αντιμετώπισης των διασυναριακών συνδέσεων και ενίσχυσης των ε, μηχανισμών μας προστασίας κατά των τραπεζικών κρίσεων. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Θα απαντήσω σε ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ κυρία Νουή. Περνάμε σε ερωτήσει. Ο κ. Μπάλτσεκ, μέρο του ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Ανουή, χαίρομαι που βρίσκεστε πάλι εδώ στην Επιτροπή μας. Έχω τρει ερωτήσεις. Καταρχάς, ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φροντίζουμε ιδιαίτερα να υπάρχει ε, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στο νομισματικό κομμάτι και το εποπτικό. η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, ε, δεσμεύτηκε να μας ε, αναφέρει και στην κατακτική φάση του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού πώς πραγματοποιείται αυτός ο διαχωρισμός. Έχουμε λοιπόν την ολοκληρωμένη αξιολόγηση, το Comprehensive Assessment, που θα πρέπει να βρίσκεται στα χέρια των εποπτών και δεν ε, θα πρέπει να δεσπόζεται από άλλους. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω από τη δική σας πλευρά πώς διασφαλίζεται αυτό ακριβώς. Δεύτερη ερώτηση. Πώς διασφαλίζεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ο ενιαίος εποπτικός μηχανισμός να μην εξαρτώνται υπερβολικά από τους εξωτερικούς συμβούλους. Οι εξωτερικοί αυτοί σύμβουλοι μπορούν να ασχοληθούν με τις ε, συστάσεις αναχώρα. Πώς κρίνετε εσείς την εμπειρογνωμοσύνη τους ε, στο θέμα αυτό και ε, τρίτον όσον αφορά την εξέταση των τραπεζών, τους ελέγχους των τραπεζών που πραγματοποιούνται. Πώς πραγματοποιούνται, πώς μπορείτε να εξηγήσετε ότι δίδεται ιδιαίτερο βάρος σε ε, μικρά στεγαστικά δάνεια, ενώ δεν ε, εξετάζονται, για παράδειγμα, για επενδύσεις σε αεροπλάνα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, κυρία Νουή. Σας ευχαριστώ όσον αφορά το διαχωρισμό ανάμεσα στην νομισματική πολιτική και την εποπτεία. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Πράγματι, θα καθοριστούν κανόνες στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και έχουν ξεκινήσει οι εργασίες πάνω στο θέμα αυτό. Είναι λεπτό το θέμα, διότι Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η αναγκαιότητα του διαχωρισμού, από την άλλη όμως να υπάρχει η δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε συνέργειες, ιδιαίτερα όσον αφορά την μακροπροληπτική εποπτεία και την χρηματοοικονομική σταθερότητα. Χάρη στον κανονισμό για τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό ε, έχει σημαντικές αρμοδιότητες και μέσα τώρα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Θα πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε να εκμεταλλευτούμε τις ε, πιθανές συνέργειες στον τομέα αυτό. Μόλις υπάρξει σχετική απόφαση, θα ενημερώσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι όμως ε, κάπως νωρίς αυτή τη στιγμή. Όσον αφορά την ολοκληρωμένη αξιολόγηση, το Comprehensive Assessment, Θέλουμε να έχουμε ισχυρό, αξιόπιστο αποτέλεσμα, έχουμε απόλυτη διαφάνεια όσον αφορά τη μεθοδολογία. Το εγχειρίδιο έχει δημοσιευτεί πρόσφατα. Έχουμε διασφάλιση της ποιότητας σε όλα τα επίπεδα, και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο Υπάρχουν επίσης ομάδες για κάθε χώρα όπου συμμετέχουν επόπτες από εθνικές εποπτικές αρχές που θα πάνε σε διάφορες χώρες για να πραγματοποιηθεί αξιολόγηση ομοτήμων για να διασφαλιστεί η ποιότητα. Επίσης φροντίζουμε να έχουμε ισχυρή διακυβέρνηση στο πρόγραμμα αυτό. Συμβουλευόμαστε το ε, ε, Διευθυντικό Συμβούλιο και σε όλες τις αποφάσεις ε, το Διευθυντικό Συμβούλιο έχει την τελευταία λέξη. Όσον αφορά ε, την επιρροή των εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, αν κατάλαβα σωστά. Ε, ιδιαίτερα αναφέρεστε στους ε, συμβούλους. Ο ε, έχει προσληφθεί με τα αποδιαδικασία που συνάδει απόλυτα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες περί δημόσιων προμηθειών. Εργάζονται οι εμπειρογνώμενες αυτοί υπό την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και έχουμε θέσει κατευθυντήριες γραμμές για τα κριτήρια επιλογής για τις 18 χώρες που χρησιμοποιούν ε, συμβούλους. Κάτι που ε, απαιτείται λόγω του μεγέθους του εγχειρήματος αυτού και για να, ε, για να υπάρχει αξιοπιστία. Εγώ λοιπόν νιώθω απόλυτα άνετα με το αποτέλεσμα οι ελεγκτές αυτοί δεν είναι αυτοί που είναι αρμόδιοι για τις τράπεζες, ούτε συμμετείχαν σε stress τεστ, σε ασκήσεις προσωμείωσης ακραίων καταστάσεων στις ε, ίδιες χώρες. Όσον αφορά την τελευταία ερώτηση, δεν είμαι σίγουρη ότι την κατάλαβα απόλυτα. Από ό,τι κατάλαβα, έχει να κάνει με τον ε, ρόλο των ε, εγγύησεων και πώς χρησιμοποιούνται οι εγγυήσεις σε περιπτώσεις ε, μικρών ε, δανείων. Αυτή τη στιγμή εκπονούμε τις αρχές για την αξιολόγηση των εγγυήσεων. Θα εφαρμόσουμε την αρχή της αναλογικότητας και θα πρέπει να γίνει η αξιολόγηση αυτή με βάση τις ίδιες αρχές σε όλες τις χώρες, ώστε να έχουμε ίσες συνθήκες ανταγωνισμού. Σας ε, ευχαριστώ πολύ. Η Ελίζα Φερέιρα, παρακαλώ. Thank Ευχαριστώ που είστε εδώ ξανά μαζί μας σήμερα. Μας φέρατε καλά νέα. Φαίνεται ότι ελέγχετε αυτό το περίπλοκο έργο που σας έχει ανατεθεί. Και ό,τι αφορά τη συνέχεια που στην Τραπεζική Ένωση, το τρίτο θέμα το οποίο θίξατε κατά κάποιο τρόπο. Είπατε ότι ε, ε, χρειάζεται ένα πολύ καλό μηχανισμό εξυγίανσης και μας δώσατε μερικά στοιχεία αυτού. Μπορείτε να μας δώσετε λίγο περισσότερες σημασίες για το πόσο σημαντικό είναι για την ποιότητα της εποπτείας ε, η ποιότητα του μηχανισμού εξυγίανσης γιατί αυτή τη στιγμή ολοκληρώνουμε τις διαπραγματεύσεις και θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι δεν δεχόμαστε μια κακή συμφωνία. Μπορείτε να μας δώσετε λίγο περισσότερες πληροφορίες γι' αυτό. Δεύτερο ερώτημά μου, η μεταβατική περίοδος για τον ενιαίο μηχανισμό εξυγίανσης. Αρχικά είχαμε τριετή περίοδο ε, προκειμένου να διευκρινιστεί τι αποτελεί ε, legacy ε, πριν περάσουμε στο καινούριο σύστημα. Μετά, πώς πιστεύετε ότι ε, η, το, ε, το ε, Συμβούλιο της Ολομέλειας θα μπορέσει να συνεργαστεί σωστά με το Εκτελεστικό Συμβούλιο έτσι ώστε οι συζητήσεις που γίνονται στο ένα να μην επαναλαμβάνονται στο άλλο. Πώς μπορεί να γίνει ο διαχωρισμός αυτών των αρμοδιοτήτων αυτών των δύο οργάνων. Θα ήθελα τη γνώμη σας. Η Ελίζα είναι η συγγήτρια για τον νέο μηχανισμό εξυγίανσης, κάνει εξαιρετική δουλειά, ε, δίνω τώρα στην κυρία Νουή. Ε, παρακολουθούμε πολύ στενά και από κοντά αυτή τη δουλειά του μηχανισμού Είναι πολύ σημαντικό γιατί ε, θέλουμε η διαδικασία, η νομοθετική διαδικασία για το μηχανισμό εξυγίανσης ε, να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό και να τεθεί σε λειτουργία ο μηχανισμός. Χρειαζόμαστε μια διαδικασία λήψη αποφάσεων αποτελεσματική γιατί η εξυγένση απαιτεί γρήγορες και αποτελεσματικές αποφάσεις. Ο χρόνος πάντα πιέζει σε τέτοιες υποθέσεις. Θα πρέπει η διαδικασία λήψη απόφαση λοιπόν να είναι όσο δυνατό πιο σύντομη. η εξυγένση θα πρέπει να ξεκινάει αν όχι μέσα στις 24 ώρες αλλά ε, σε ένα Σαββατοκύριακο. Σε ό,τι αφορά το ενιαίο Ταμείο Εξυγένσης, δεδομένου ότι ε, ο ευρωπαϊκός τραπεζικός τομέας θα πληγεί όσο ε, παραμένουν οι εθνικοί μηχανισμοί. Οπότε τα 10 χρόνια είναι υπερβολικά μακρά περίοδος. Ε, ίσως θα πρέπει να μειωθούμε στα και ακόμα καλύτερα, να το μειώσουμε στα 5 και ακόμα καλύτερα στα 3 χρόνια. Αυτό δεν απαιτεί διπλασιασμό των εθνικών συνεισφορών, οι οποίες μπορούν να ε, έχουν καταβληθεί μετά από μια συγκεκριμένη περίοδο χρόνου. Ε, από εκεί και πέρα το ταμείο θα είναι κοινό ευρωπαϊκό. Ε, τώρα, ε, χρειαζόμαστε προστατευτικό μηχανισμό και για την προσωρινή μεταβατική περίοδο και για τη μόνιμη περίοδο. Ο, το ενιαίο ταμείο θα πρέπει να έχει δυνατότητα δανεισμού, όπως προβλέπεται και από το μηχανισμό εξυγένσης. Ο, ο, προστατευτικός, ο κοινός προστατευτικός μηχανισμός, ήδη από τη μεταβατική περίοδο, είναι απαραίτητος για να ε, ε τον ίδιο τρόπο όλες τις δεδομένου ότι από τις πρώτες περιόδους, από τις πρώτες υποθέσεις εξηγένσης μπορεί να εκμηδενιστούν, να, ε, να εξαφανιστούν τα ε, ποσά που διαθέτει ο μηχανισμός. Το οποίο σημαίνει ότι χρειαζόμαστε, θα αν δεν έχουμε ευρωπαϊκό μηχανισμό προστασίας, θα χρειάζεται να έχουμε πολλούς εθνικούς μηχανισμούς ε, προστασίας. Χρειαζόμαστε όμως τον ευρωπαϊκό μηχανισμό για να εξασφαλίσουμε την ίδια μεταχείριση σε όλες τις τράπεζες τις οποίες θα εξηγιανθούν. Ο, ο μηχανισμός αυτός θα, ε, θα χρηματοδοτείται από όλες τις τράπεζες και όχι μόνο από τις τράπεζες οι οποίες είναι υπό εξηγίαση. Θα πρέπει να είναι δηλαδή πραγματικά ευρωπαϊκός αυτός ο μηχανισμός. Σε ό,τι αφορά το θέμα της μεταβατικής περίοδου. Ε, τα πράγματα θα διευκρινιστούν μετά το, τη λήξη του, της ε, συνολικής αξιολόγησης. Θα εντοπίσουμε τα ε, χαρτοφυλάκια που είναι τα πιο ε, δημιουργούν τους περισσότερους κινδύνους, τα πιο αδιαφανή, αυτά τα οποία μάλλον θα εντοπίσουμε τα μη χρηματοδοτούμενα δάνεια, ε, όλα αυτά θα τα ξέρουμε στο τέλος της διαδικασίας αξιολόγησης. Μετά από αυτή την αξιολόγηση θα ε, εντοπιστούν οι, ε, οι αδυναμίες, οι, οι ελλείψεις ε, πιστώσεων η έλλειψη κάλυψης και ε, θα προσφύγουμε στους, ε, στον Εθνικό Μηχανισμό, Προστατευτικό Μηχανισμό και κατόπιν στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό ε, του Εξυγίανσης για την ανακεφαλαιοποίηση ενδεχομένως της τράπεζας. Όμως όλα αυτά θα γίνουν σαφή στο τέλος της διαδικασίας αξιολόγησης. Σε ό,τι αφορά την κατανομή αρμοδιοτήτων και εξουσιών ανάμεσα στην, ε, στο ε, Συμβούλιο Ολομέλειας και στο Εκτελεστικό Συμβούλιο. Δεν γνωρίζω πολύ καλά τις λεπτομέρειες για να σας απαντήσω. Αλλά το Εκτελεστικό Συμβούλιο προφανώς θα πρέπει να έχει πραγματικές ισχυρές εξουσίες για να πάρει τις αποφάσεις. Προφανώς βέβαια θα πρέπει να είναι υπόλογο προς το ε, ε, Συμβούλιο Εξ, ε, της Ολομέλειας και στα ευρωπαϊκά όργανα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος του Θα ήθελα να σας κάνω δύο ερωτήσεις. Πρώτον, δεν θέλουμε ο νέος εποπτικός μηχανισμός ε, να κάνει διαχωρισμό μεταξύ της Ευρωζώνης και της υπόλοιπης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε λοιπόν τα μέλη τα κράτη-μέλη που δεν είναι μέλη της Ευρωζώνης να συμμετάσχουν το ταχύτερο δυνατόν στον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό τι πρέπει να γίνει και τι πιστεύετε ότι θα μπορούσε να γίνει και πώς θα πρέπει να αναλάβει την επιτάχυνση αυτής της διαδικασίας. Να πείσουμε δηλαδή τα κράτη που δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη να συμμετάσχουν εθελοντικά στο SSM. Το δεύτερο αφορά τον έλεγχο ποιότητας δεδομένων των χρονικών περιορισμών. Σαφώς θα πρέπει να βασιστείτε στην υποστήριξη των ε, εμπειρογνωμόνων εξωτερικών. Γνωρίζουμε όλοι ότι αυτοί οι εμπειρογνώμονες ε, δεν κάνουν πάντα καλή δουλειά όπως έχουμε διαπιστώσει στο παρελθόν. Πώς θα διασφαλίσετε λοιπόν ότι η ποιότητα των υπηρεσιών αυτών των εμπειρογνωμόνων θα είναι η κατάλληλη για το έργο αυτό, για το εγχείρημα. Ευχαριστώ. Σύμφωνα απόλυτα μαζί σας, δεν πρέπει να υπάρξει διαχωρισμός μεταξύ χωρών της Ευρωζώνης και χωρών εκτός Ευρωζώνης. Δύο είναι οι τρόποι για να διασφαλίσουμε ότι αυτό δεν θα συμβεί. Ο πρώτος είναι να συνεργαστούμε στενά με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τραπεζών, την EBA, που έχει αναλάβει το Single Rule Book, το ενίο βιβλίο κανονών, και για παράδειγμα τα περισσότερα εργαλεία για τον ελεγχό της ποιότητας του ενεργητικού και για τα ποιοτικά stress προέρχονται από την ΕΜΠΑ. Εγώ είμαι πεπισμένη ότι η συνεργασία μεταξύ των χωρών που θα ανήκουν στο SSM και των χωρών που δεν θα ανήκουν είναι ένα θέμα που εγώ υπερασπίζομαι προσωπικά. Φροντίζω να συμβαίνει. Θέλω να φροντίσουμε να συμβαίνει και στο μέλλον επί όλων των ε, σημείων, όλων των στοιχείων. Εγώ προσφέρθηκα εθελοντικά ενώπιον του Εποπτικού Συμβουλίου να είμαι μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τραπεζών, της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, της EBA. Παρά του μεγάλου φόρτου εργασία που έχω στη Φραγκφούρτη, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η σχέση λοιπόν με την ΣΕΒΑ είναι πολύ σημαντική. Όσον αφορά την εθελοντική συμμετοχή των χωρών που δεν ανήκουν στο SSM, στο SSM ελπίζω να συμβεί. Για να διασφαλίσουμε κάτι τέτοιο, το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να κάνουμε πολύ καλή δουλειά και έχουμε δεσμευτεί για κάτι τέτοιο όσον αφορά την εποπτεία στον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό. Συγγνώμη, δεν απάντησα στη δεύτερη ερώτηση που αφορά τη διακυβέρνηση της ολοκληρωμένης αξιολόγησης ε, όσον αφορά τη χρήση εμπειρογνωμόνων εξωτερικών ελεγκτών. Συζητήσεις γίνονται σε διάφορα επίπεδα για τη συμμετοχή, τη συνεργασία, την διακυβέρνηση, την παροχή συμβουλών, τους οικονομικούς ελέγχους. Έχουμε έναν επικεφαλής έργου, τον Τζούκα Βεζαλά, από την Γενική Διεύθυνση Macroprudential αριθμός 3. Επίσης ε, έχουμε μια διοικητική επιτροπή της ολοκληρωμένης αξιολόγησης όπου μπορούν να αμφισβητηθούν οι προτάσεις των συμβούλων και των ελεγκτών. Έχουμε ένα κεντρικό γραφείο ολοκληρωμένης αξιολόγησης όπου προετοιμάζονται και εξετάζονται μεθοδολογίες επίσης. Έχουμε εθνικά γραφεία για την ολοκληρωμένη αξιολόγηση σε όλες τις εθνικές αρμόδιες αρχές. Φυσικά συμβουλευόμαστε τις εθνικές ε, αρμόδιες αρχές πριν προχωρήσουμε με τη μεθοδολογία. Εξετάζουμε ε, με κριτικό πνεύμα τις προτάσεις, με στενών διαλόγων, με τις τράπεζες, τις ε, Ομοσπονδίες Τραπεζών, τις Ομοσπονδίες Οικονομικών Ελεγκτών σε τακτική βάση. Είμαι λοιπόν ε, βέβαιη ότι η διακυβέρνηση είναι όσο καλή θα μπορούσε να είναι σε αυτό το εγχείρημα. Ευχαριστώ κύριε Νοή εκ μέρους του ECR, ο κύριος Σιλέ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Νοή για την ε, πολύ ολοκληρωμένη εισαγωγή σας. Έχω δύο ερωτήσεις. Η μία σχετίζεται με την επίσημη συνεργασία ανάμεσα στον εποπτικό μηχανισμό ή το εποπτικό συμβούλιο με ε, τις Ηνωμένε Πολιτείες, τον Καναδά και άλλες χώρες ε, με τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ήδη να έχει συμφωνίες εμπορίου και επενδύσεων ή με τις οποίες ε, θα ε, συνάψει τέτοιες συμφωνίες. Ε, έχουν να κάνουν λοιπόν με συμφωνίες για την είσοδο στην ευρωπαϊκή αγορά και έτσι υπάρχει ενδεχομένως συστηματικός κίνδυνος, συστημικός κίνδυνος για την ευρωπαϊκή αγορά. Και η δεύτερη μερότηση ερώτηση σχετίζεται με αυτό που ρώτησε ο Βολφ Κλίνς. Έχει να κάνει με τις τράπεζες εκτός Ευρωζώνης που λειτουργούν εντός της Ευρωζώνης όπως ε, η Σουηδική Τράπεζα, η οποία τεσπόζει στην αγορά των βαλτικών κρατών. Ε, σύντομα περιμένουμε όλα τα κράτη της Βαλτικής ε, να εισέλθουν στη ζώνη του ευρώ, προς τη μήνυνη είναι δύο. Πώς θα μπορείτε λοιπόν αποτελεσματικά να εποπτεύετε τις τράπεζες αυτές. και η εποπτεία αυτή θα ισχύει και για τις μητρικές τράπεζες που βρίσκονται εκτός της ζώνης του ευρώ. Σας ευχαριστώ. Πράγματι, συνομιλούμε πολύ με ε, ε, θεσμούς εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σχετικά με την ολοκληρωμένη αξιολόγηση. Πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο να εξηγούμε τι κάνουμε, να επιδείξουμε τη βούλησή μας να είμαστε απολύτως διαφανείς όσον αφορά το περιεχόμενο και τη μεθοδολογία του εγχειρήματος αυτού για να αποκαταστήσουμε την ε, εμπιστοσύνη προς τις Ευρωπαϊκές Τράπεζες. Μάλλον θα προσέξατε ότι είμαστε μία ότι ένας από τους τέσσερις ε, γενικούς διευθυντής ήταν ε, παλαιότερα Αμερικανός επόπτης. Μπορούμε λοιπόν να μάθουμε από αυτόν και είμαι πολύ περήφανη που ένας ε, από τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ε, θα είναι επόπτης από τον Καναδά που ακόμα ελέγχει τράπεζες εκεί. Αυτός λοιπόν είναι ένας άλλος τρόπος να μάθουμε από άλλους οργανισμούς και να εφαρμόσουμε τις ε, καλύτερες πρακτικές. Όσον αφορά τις μη ευρωπαϊκές τράπεζες ε, στην ζώνη του ευρώ, οι τράπεζες που δεν εμπίπτουν ε, στον ενιαίο υποπτικά μηχανισμό, τους τελευταίους τρεις μήνες έχουμε επικεντρωθεί πάρα πολύ στις σχέσεις αυτές. Τέλη Ιανουαρίου είχαμε ένα σεμινάριο για τους ε, επόπτες των θηγατρικών που δραστηριοποιούνται ε, εκτός ε, του ενιού εποπτικού μηχανισμού. Κάποιες, από, κάποιες χώρες έστειλαν εκπροσώπους και στα δύο αυτά σεμινάρια Πιστεύω λοιπόν ότι έχουμε βρει την σωστή ρύθμιση. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Θα συνεχίσουμε να καταβάλουμε προσπάθειες για να βρούμε τον καλύτερο μηχανισμό όσον αφορά την εποπτεία των τραπεζών του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού όσον αφορά τις σκανδιναβικές ρυθμίσεις. Ε, εκτιμώ ιδιαίτερα τα όσα έχουν γίνει στο, στην περιοχή αυτή. Ζήτησα από τους συνεργάτες μου να μου εκπονήσουν ε, ένα έγγραφο σχετικά με τις σκανδιναβικές ρυθμίσεις και έχουμε υιοθετήσει κάποιες ιδέες από αυτές. Μεταξύ άλλων ε, τις ε, κοινέ επιτόπου έρευνες. Θα φροντίσουμε λοιπόν αυτές οι βέλτιστες εποπτικές πρακτικές να ακολουθούνται. αρμόδιος ε, για την ε, σύνταξη του ε, εγχειριδίου για την εποπτεία, προέρχεται από την Φιλανδία, γνωρίζει πολύ καλά λοιπόν τις σκανδιναβικές ρυθμίσεις και θα φροντίσει όχι μόνο να μην δημιουργηθούν δυσκολίες, αλλά ε, για καλύτερη ένταξη των ε, χωρών εκτός ε, Ευρωζώνης στις ρυθμίσεις του ενιαίου υποπτικού μηχανισμού. Ευχαριστώ κύριο Σεγκίκολτ. Καλώς ήρθατε κυρία Γκίκολτ στην Επιτροπή μας. Δύο ερωτήσεις έχω. Η πρώτη έχει να κάνει με τις παρατηρήσεις σας και αυτές που κάνετε εδώ προφορικά αλλά και στις γραπτές σας απαντήσεις για τις οποίες σας ευχαριστώ. Είπατε ότι το Εποπτικό Συμβούλιο σκοπεύει να μας στέλνει πρακτικά των διαδικασιών σε τριμηνία βάση. Στις ε, μακροσκελείς διαπραγματεύσεις, η Σιλβί ο ε, θα θυμούνται τις διαπραγματεύσεις αυτές. Στις διαπραγματεύσεις αυτές λοιπόν ε, ζητήσαμε κάτι που να μοιάζει πρακτικά. Με πρακτικά. Δεν χρησιμοποίησαμε τη λέξη πρακτικά για να μην δημιουργήσουμε προηγούμενο για τα όσα συμβαίνουν ε, στο, στο Διευθυντικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ε, στην περίπτωση αυτή όμως θέλαμε να βρούμε έναν αντίστοιχο όρο και γι' αυτό οι πληροφορίες αυτές ε, θα πρέπει να μας αποστέλλονται μετά την πραγματοποίηση των συναντήσεων. Είπατε λοιπόν ότι είσαστε διατεθειμένοι να μας στείλετε το υλικό αυτό και θα σας παρακαλούσα να τηρήσετε αυτά που συζητήσαμε στο πλαίσιο του μηχανισμού. Και επίσης θα ήθελα να αναφερθώ στην ερώτηση του Wolf Klins. Είσαστε διατεθειμένοι να μας δώσετε έναν κατάλογο με τους συμβούλους και σε ποιες τράπεζες εργάζονται. Είδαμε κάποια ονόματα στον ε, οικονομικό τύπο. Θα ήταν όμως μια διαφανής διαδικασία να μοιραστείτε μαζί μας ε, τα ονόματα των ε, οικονομικών συμβούλων και σε ποιες τράπεζες εργάζονται. Θα ήταν δυνατό να το κάνετε αυτό. Κύριε Νούη, σε ό,τι αφορά τα πεπραγμένα, κάτι που να μοιάζει με πρακτικά, έτσι και εμείς το καταλάβω, έχουμε καταλάβει, δεν υπάρχει διαφορά σε αυτό μεταξύ μας. Σημειώνω ότι ζητάτε μετά τις συνεδρίασης να γίνεται μια τέτοιου τύπου ενημέρωση, όχι κάθε τρίμηνο. Ε, για μας το τρίμηνο φαινόταν λογικό όταν ελήφθη η απόφαση, αλλά θα ενημερώσω το Διοικητικό Συμβούλιο, το Εκθεστικό Συμβούλιο και νομίζω δεν θα έχουν αντίρρηση. Σε ό,τι αφορά τον κατάλογο του ποιοι συμβούλοι δουλεύουν για κάθε τράπεζα, για ποιες τράπεζες. Δεν μπορώ να απαντήσω σήμερα, σας υπόσχομαι θα απαντήσω αργότερα. Θέλω να ρωτήσω αν από νομικής πλευράς μου επιτρέπεται να δώσω απάντηση. Γιατί ορισμένοι σύμβουλοι και εξωτερικοί και δικοί μας σύμβουλοι ε, ε, προσελήφθησαν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά οι υπόλοιποι είναι από εθνικές αρχές, οπότε πρέπει να ρωτήσω να δω αν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Ε, θα ήθελα μια δεύτερη ερώτηση για το ίδιο θέμα. Σε ευχαριστώ πολύ που θα το εξετάσετε. Ε, καταλαβαίνω τη διαφορά μεταξύ των δύο αυτών ομάδων συμβούλων, αλλά θα μας έδινε κάποιες απαντήσεις γιατί τα ονόματα που είδαμε στον οικονομικό τύπο ε, μας άφηναν να, ε, άφηναν να διαφανεί ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Ορισμένοι από τους ε, συμβούλους έλεγξαν μια τράπεζα από μερικά χρόνια, τώρα ανέλαβαν, μετά ανέλαβαν, συγγνώμη, δούλευαν για μια τράπεζα πριν μερικά χρόνια και μετά έγιναν σύμβουλοι που θα ελέγξουν την ίδια τράπεζα. Οπότε είναι δύσκολο να κάνουν καλά το καθήκον τους. Ε, οπότε θα ήθελα να ρωτήσω πώς διαχειρίζεστε αυτές τις ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων τη στιγμή της επιλογής των συμβούλων σας. Απάντηση. Πράγματι, οι εταιρείες ελεγκτών είναι περιορισμένες σε αριθμό. Εμείς ε, στα κριτήρια τα οποία δώσαμε ως Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις εθνικές ε, εποπτικές αρχές ήταν να μην χρησιμοποιηθούν ελεγκτές που έχουν έρθει σε επαφή με την τράπεζα τα τελευταία δύο οικονομικά έτη. Δεν είναι και πολύ μεγάλη περίοδο, το αναγνωρίζω, αλλά αυτό ήταν το κριτήριο το οποίο έδωσε η, η, η προπόθεση που έδωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Οπότε ενδεχομένω Προσελήθηκαν κάποιοι ελεγκτές που δεν είχαν επαφή με τις συγκεκριμένες τράπεζες τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά πριν από τρία χρόνια. Ευχαριστώ για μέρος του ΕΛΚ, κ. Ντόρτμαν. Ευχαριστώ κυρία Νόη που βρίσκεστε εδώ. Στη... Επικρίναμε πρόσφατα το Ιταλικό τραπεζικό σύστημα και ειδικότερα τις μικρές Ιταλικές τράπεζες υπόθηκε κατακριματισμός, αναφέρθηκε κατακριματισμός του τραπεζικού τομέα ε, στην Ιταλία με υψηλό τραπεζικό δίκτυο, χαμηλή κερδο... κερδοφορία και αναφέρθηκε ότι οι συνεταιριστικές τράπεζες ε, στην Ιταλία είναι ο αδύναμος κρίκος του Ιταλικού τραπεζικού συστήματος. Αν δείτε τι συμβαίνει πραγματικά επί τόπου και εγώ έρχομαι από μια περιοχή που έχουμε πολλές μικρές συνεταιριστικές τράπεζες πρέπει να πω ότι αυτές οι συνεταιριστικές τράπεζες τα τελευταία χρόνια απλά έκαναν το καθήκον τους. Έδωσαν πιστώσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πιστώσεις σε οικογένειες, απέφυγαν το capital crunch έχουν 14% ε, κεφάλαια ε, κατηγορία 1. Μου φαίνεται λοιπόν περίεργο αυτό που είπε ο Επίτροπος Ρέν για τις τράπεζες αυτές. Έχετε εσείς κάποια άποψη γι' αυτό και ποια είναι αυτή. Δεν θα, αναφέρω ένα, δεν θα αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο τραπεζικό σύστημα αλλά να πω ότι στην Ευρώπη υπάρχει περιθώριο για πολλά διαφορετικά επιχειρηματικά μοντέλα στις τράπεζες. Μικρές τράπεζες, μεσαίες, μεγάλες, διεθνείς και μονοεγχώριες ε, λιανικών υπηρεσιών και τραπεζές που ασχολούνται με μεγάλες επιχειρήσεις. Δεν πιστεύω λοιπόν ότι η υγεία μιας τράπεζας ε, βασίζεται στο μέγεθος, στο ε, ε, ε, επιχειρηματικό μοντέλο βάσει το οποίο λειτουργεί. Κατά την απόψή μου, οι τράπεζες που πρέπει να πάψουν να υπάρχουν είναι αυτές που ο Μάριο Τράγκη ονόμασε τράπεζες ζόμπι που είναι υπερφορτωμένες με υπερβολικά μη εξυπηρετούμενα στοιχεία ενεργητικού ό,τι μορφή και αν έχουν αυτά. Γι' αυτό το λόγο δεν μπορούν να παράσχουν δάλια στην οικονομία. Αυτές προσπαθούμε να εντοπίσουμε στην ολοκληρωμένη αξιολόγηση και ελπίζω ότι μετά από αυτή την αξιολόγηση θα αναλυθούν οι απαραίτητες δράσεις ώστε να πάψουν να υπάρχουν αυτές οι τράπεζες ζόμπι. Ευχαριστώ κύριε Τώρα εκ μέρου τη κυρία Τάισεν. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη, διότι ήθελα να παρευρίσκεται, αλλά λόγω απρόπτων ε, συνθήκων δεν μπόρεσε να βρίσκεται εδώ σήμερα. Ζητάει συγγνώμη, λοιπόν. Δίνω τώρα το λόγο στον Αντολίν και ο Σάντσες Ευχαριστώ. τρει ερωτήσει. Πρώτον, ε, πώς προβλέπετε η μετάβαση ε, το σύστημα θα αρχίσει να λειτουργεί πλήρως από τον Νοέμβρη και μετά, οπότε μέχρι τότε έχουμε μια μετάβαση. Τι έχει προβλεφθεί για αυτή την περίοδο. Για να αποφύγουμε αλληλεπικαλύψεις στην εποπτεία. Δεύτερον, για το πλαίσιο του financial reporting. Τι έχει προβλεφθεί και πάλι για να αποφύγουμε την αλληλεπικάλυψη εκθέσεων και για να ε, μην προκύψει βομβαρδισμός πληροφοριών για μη σημαντικά θέματα. Τρίτον, ενημερωθήκαμε για το ότι έγινε ε, μια αξιολόγηση της Βασιλείας 3. Ε, περιέλαβε 202 ιδρύματα και από ό,τι φάνηκε ότι δεν έχουν περισσότερα προβλήματα από τα υπόλοιπα ιδρύματα. Αυτό οδήγησε το συμπέρασμα ότι δεν θα πρέπει να ε, οδηγηθούμε σε πιο ευρία έρευνα και άλλων φορέων σε σχέση με τα Βασιλεία 3. Μπορείτε να μας σχολιάσετε. Thank you. Ε, Ευχαριστώ. Σε ό,τι φορά τη μεταβατική περίοδο, το κατά πόσο θα είμαστε έτοιμοι το Νοέμβριο για να ξεκινήσουμε την, ως ευρωπαϊκός μηχανισμός, εποπτικός μηχανισμός. Ναι, η απάντηση είναι ρητά ναι. Ε, είμαστε, τηρούμε το χρονοδιαγράμμά μας ε, σε όλα τα μέτωπα. Έχουμε θέσει προτεραιότητες σε ό,τι αφορά τα καθήκοντά μας. Έχουμε διακρίνει δηλαδή μεταξύ αυτών που είναι απολύτως απαραίτητα και γρήγορα και αυτών τα οποία ε, θα ήταν καλό να τα έχουμε μέχρι τον Νοέμβρη αλλά μπορούν και να αναβληθούν. Είμαι απόλυτα πεπισμένη ότι είναι δυνατόν όλα αυτά να γίνουν έγκαιρα με αξιόπιστο τρόπο. Επίσης, ε, έχουμε σκεφτεί και την μεταβατική περίοδο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου. συζητούμε με τις Εθνικές Εποπτικές Αρχές προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουν πάρει πριν από τον Νοέμβρη τις ε, απαραίτητες αποφάσεις προκειμένου ε, να μην, δημιουργηθούν, να μην δημιουργηθεί σύγχυση τη στιγμή της μετάβασης. Νομίζω ότι είμαστε σε καλή κατάσταση, σε καλό στάδιο και σε αυτό το επίπεδο. Είπατε να μην υπάρξει αλληλεπικάλυψη στην εποπτεία. Ναι, αυτός είναι ο στόχος. Νομίζω ότι ο κανονισμός κάνει σαφή διάκριση ανάμεσα στις σημαντικές και στις λιγότερο σημαντικές τράπεζες. Παρ' όλα αυτά το σύστημα είναι ενιαίο, με, ενιαία, με ενιαίους ε, κανόνες και συστάσεις για την εποπτεία που θα εφαρμόζονται σε όλες τις ευρωπαϊκές τράπεζες ε, του ε, μηχανισμού. Οπότε έτσι περνάω και στην ερώτηση σχετική με το reporting, με την υποβολή εκθέσεων. Αναγνωρίζω ότι αυτή τη στιγμή για την συνολική αξιολόγηση συλλέγουμε πολλές πληροφορίες, πολλά δεδομένα. Αλλά αυτό γίνεται προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι θα ε, να εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή αξιοπιστία για τις ευρωπαϊκές τράπεζες. Σε ό,τι αφορά τις μελλοντικέ αναφορές θα συλλέγουμε τις εκθέσεις για τα δεδομένα όλων των εποπτευόμενων τραπεζών, σημαντικών και λιγότερο σημαντικών, ε, ε όλα αυτά, τα περισσότερα από αυτά τα δεδομένα θα βασίζονται στις τεχνικές προδιαθέσεις της CBA Ε, η ΕΚΤ ε, θα προβλέψει να και κάποιες πρόσθετες υποχρεώσεις ε, μετά από διαβούλευση, εντάξει, κάτι πρόσθετο του EBA, της EBA, της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τραπεζών, γιατί μπορεί να υπάρξουν πρόσθετες ανάγκες. Επίσης θα χρειαστούμε ε, και, σε, και, τις, ε, ε, και κάποιες πρόσθετες πληροφορίες σε ό,τι αφορά τις, τους ισολογισμούς των τραπεζών Τώρα εκεί θα έχουμε διάκριση ανάμεσα στις πιο σημαντικές και λιγότερο σημαντικές ε, τράπεζες. Για τις, πιο, για τις λιγότερο σημαντικές τράπεζες θα προσπαθήσουμε να μην ζητάμε ε, πάρα πολλά, υπερβολικά πολλά από αυτές που είναι μικρές τράπεζες κατά βάση. Θα υπάρχει δηλαδή ένα κατόφλι. Ε, ούτε υπάρχει υποχρέωση χρήσης του διεθνούς προτύπου χρηματοοικονομικής αναφοράς του IFRS. από αυτές τις τράπεζες. Δηλαδή οι απαιτήσει για τις μικρές τράπεζες, τα μικρά ιδρύματα είναι αναλογικές με τις, σε αναλογία με τις δυνατότητές τους. Ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος στην κυρία Γκουλάκ. Καλημέρα κύριε Νούη. Ευχαριστούμε που βρίσκετε μαζί μας όπως επιθυμούσαμε και χαιρόμαστε που σας βλέπουμε εδώ. Εγώ έχω μια ερώτηση που μοιάζει με τις ανησυχίες της Λίζα για το ψήφισμα. Ε, και εγώ συμμετείχα ως ε, σκιώδης είναι ένα βασικό ερώτημα, όχι τεχνικό. Δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει ότι θα θέλαμε να κλείσουμε γρήγορα συμφωνία, ενώ επί της ουσίας δεν γνωρίζουμε πώς ε, υπολογίζονται οι συμβολές των τραπεζών. Αυτό μου δημιουργεί καταρχάς δημοκρατικό πρόβλημα και δεν ξέρουμε αν θα πρέπει να εντάσσεται σε πράξη του Συμβουλίου ή σε τη πράξη, αλλά υπάρχει και κάτι άλλο που ανησυχεί. Μιλάμε για πολύ υψηλά ποσά. που μπορούν να δημιουργήσουν διαστρεβλώσεις ε, στην εκάστοτε χώρα λόγω τη ε, διαφορετική μορφή των τραπεζικών συστημάτων. Και εν τέλει, εγώ αναρωτιέμαι πω αυτό θα έπρεπε να εμβαθύνουμε περισσότερο πριν καταλήξουμε σε συμφωνία. Διότι αν ε, πούμε ότι υπάρχει ε, εξυγίανση και υπάρχει ένα ταμείο και δεν ξέρουμε ποιο έχει πρόσβαση σε αυτό και πώ, και αυτό έχει συνέπειε για τα δημοσιοοικονομικά, όπου μεγάλη οι ε, τραπεζικοί όμιλοι σε κάποιες χώρες θα χάσουν πολλά χρήματα και ελπίζω ότι η Γενική Διευθύνση Εκφήνη δεν θα έρθει να τους πει ότι αυτό θα ε, χρεωθεί τελικά στον προπολογισμό του κρατικού. Δηλαδή σε τελική ανάλυση πάλι οι φορολογούμενοι θα πληρώσουν. Διότι μειώνεται σημαντικά ο φόρος ε, προς τις επιχειρήσεις. Και αναρωτιέμαι πως εκεί η προσέγγιση παρεκκλίνει. Είναι πολιτικά τα ζητήματα, αλλά Μήπως το σύστημα θα έπρεπε να παγιωθεί καλύτερα ώστε τη στιγμή ενεργοποίησης του να μην ρίψουν κινδυνευτεί το σύνολο των επιχειρήσεων. Ευχαριστώ. Θεωρώ ότι πράγματι είναι πολύ σημαντικό το σημείο αυτό. Οι επόπτες έχουν επικεντρωθεί στα απαραίτητα εργαλεία, στη διακυβέρνηση, στον τρόπο λήψης αποφάσεων στον μηχανισμό εξυγένσης, στον νέο μηχανισμό εξυγένσης, στον SRM, γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο κομμάτι, όχι η φορολογία. Δεν είναι ο χώρο στον οποίο κινούνται συνήθω. Αλλά συμφωνώ, ναι, ο υπολογισμό των συμβολών των συνεισφορών πρέπει να εμβαθυνθεί. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να εξετάσουμε το πρόβλημα αυτό σε κάποιο άλλο κείμενο ώστε να μην καθυστερήσει το, το SRM και να έλθει σε ύπαρξη σε αυτή την θητεία. Νομίζω σήμερα το πρωί υπάρχει ένα άρθρο στο Financial Times το οποίο διάβαζα πριν έρθω εδώ. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να υπάρξουν σημαντικές διαστρεβλώσεις ε, ανάλογα με τη χώρα και πρέπει οπωσδήποτε να μελετηθεί το θέμα αυτό. Ναι, πολύ γρήγορα, κατά την απόψή σας, έχει νόημα να έχουμε μία τέτοια αρχή παρότι θα υπάρχει αυτή η δαμόκλειο σπάθη, δεν ξέρουμε αν θα καταφέρουν να συμφωνήσουν τα κράτη μέλη όσον αφορά τη συνεισφορά. Βλέπω, γνωρίζετε πολύ καλά τα συνταγματικά θέματα. Πιστεύω ότι πράγματι κάθε βήμα αξίζει τον κόπο, εφόσον μπορούμε να πούμε ότι θα υλοποιηθεί υπό τον όρο ότι θα υπάρχει ένα κείμενο το οποίο θα έχει εμβαθύνει σε αυτά τα ζητήματα υπολογισμού των συνεισφορών βάσει του οποίο δηλαδή θα έχει διασφαλιστεί ένα κομμάτι του SRM. Και έτσι θα έχουμε ορίσει και τις προσπάθειες που απομένουν να γίνουν ώστε να καταλήξουμε σε ένα δίκαιο και σταθερό καθεστώς ε, συνεισφορών. Γιατί πράγματι έχετε δίκιο. Εάν τη θα ενεργοποιηθούν οι συνεισφορές ε, ξαφνικά επαναστατήσουν οι πιθανοί οι φορολογούμενοι βρίσκεται σε στη θέση όλο το σύστημα ξαφνικά που δυναμώνεται. Δεν μπορούμε να πάρουμε τέτοιο κίνδυνο. Πρέπει να σταθεροποιήσουμε και να παγιώσουμε ότι υπάρχει ήδη, επειδή έχει ζητηθεί ήδη σε βάθο εδώ και μήνε, ε, για να μην πω χρόνια, και πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι για το Σούμπιο που αναφέρετε εσεί, οι εργασίε δεν έχουν βαθυνθεί ίσω ε, επαρκώ, χρειάζονται μελέτε ε, επιπτώσεων. Θα μπορούσαμε λοιπόν να προχωρήσουμε στο πρώτο σημείο, υπό τον όρο θα βρούμε μια λύση σε αυτό το πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε ολοκληρώσει τις παρεμβάσεις. Αν υπάρχει κάποιο άλλο μέλος, όπως ο κύριος Λάμπερτ, παραδείγμα, έχετε τον λόγο, κύριε Φιλίπ. Ναι, καλημέρα κυρία Ανουή. Καλώς ορίσατε. Είστε ήδη παλιά φίλοι της Επιτροπής ΕΚΟΝ. Σας βλέπουμε πολύ εδώ και αυτό είναι καλό. Παρέλθω στη σύγκρουση συμφερόντων. Διαβάζοντας ε, ένα άρθρο εδώ των Financial Times ε, ανησυχώ διότι λέει ότι όλοι μου εμάνει η εταιρεία που επιλέξει το σύμβουλο για την υλοποίηση του SSM και της ολοκληρωμένης αξιολόγησης είναι η ίδια εταιρεία που λέει στη Βρετανική κυβέρνηση προσοχή λόγω της Τραπεζικής Ένωσης η ΣΥΤ του Λονδίνου βρίσκεται σε κίνδυνο διότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, προτίθεται να δώσει κίνητρα σε κάποιες ε, τράπεζες που εποπτεύει να επαναπατρίσουν ε, τις συναλλαγές τους εντός των ορίων της Ευρωζώνης. Και η ερώτησή μου είναι, ήταν αναγκαίο να χρησιμοποιηθούν αυτοί οι οποίοι φυσικά ε, εποφελούνται από διάφορες διαφορετικές περιπτώσεις και υποθέσεις. Δεδομένου ότι είναι πολιτικά ευαίσθητο ζήτημα, ίσω να μην ήταν και η καλύτερη ιδέα να συνεργαστείτε με τέτοιου ανθρώπου οι οποίοι στο παρελθόν ε, έχουν και συμμετάσχει και σε λίγο πιο μελανές στιγμές της οικονομικής ιστορίας της Ένωσης. Η ερώτηση που θέτε είναι σημαντική. Δεν είμαι βέβαιο ότι είχαμε άλλη επιλογή. Όταν επελέγει η Όλιβε δεν υπήρχε επόπτης ε, εντός της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Χρειαζόταν λοιπόν υποστήριξη από μια ομάδα που δημιουργήθηκε από ανθρώπους που έρχονταν από την Γενική Διευθύνση Οικονομικής Σταθερότητας και από αποσπασμένα άτομα από τις, ε, ε, αρχές, ε, τις ελεκτικές αρχές της καταγωγής τους. Εδώ μιλάμε για επαγγελματίες οι οποίοι ήταν απολύτως αναγκαίο να υπάρχουν για μια τέτοια άσκηση. Αυτό που με καθησυχάζει είναι ότι διαπίστωσα ότι ο Λιβερμαν επελέγει μετά από διαγωνισμό, από πρόσκληση για υποβολή προσφορών, ανταποκρινόμενοι στις πιο αυστηρέ προδιαγραφές. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πάντα εξετάζει πολύ προσεκτικά τα θέματα αυτά. Θεωρώ λοιπόν ότι έγινε ό,τι ήταν δυνατόν ώστε οι κανόνες δεοντολογίας να τηρηθούν στο μέγιστο βαθμό. Τώρα αυτά που γράφουν οι εφημερίδες και κατά πόσο θα είναι κατάλληλη η επιλογή της Wiman Δεν έχω άποψη εγώ για το συζήτημα. Εγώ βλέπω τα άτομα που δουλεύουν μαζί μας πολλές φορές την εβδομάδα και σας διαβεβαιώ ότι είναι εξαιρετικά επαγγελματίε που ανταποκρίνονται στα αιτήματα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ηγείται του έργου αυτού παρότι βασίζεται σε συμβούλους για ένα κομμάτι μεθοδολογίας. Ε, συγγνώμη, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι αυτοί οι άνθρωποι, εδώ μιλάμε για ένα συνικό τείχος ουσιαστικά, δεν σας κάνει εντύπωση ότι ο Λίβε Γουαϊμάν που λαμβάνει λες από το κύριο Λόμπι του City του Λονδίνου προειδοποιεί τη City του Λονδίνου και τις Βρετανικές Αρχές ότι υπάρχει πρόθεση επαναπατρισμού ε, δηλαδή να δώσει κίνητρα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για επαναπατρισμό κεφαλαίων από τράπεζε τη Ευρωζώνης. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχουν τέτοια όρια σαν αυτά που λέτε και δεν πιστεύω ότι είναι αφελέ να λέμε ότι δεν θα έχουν πρόσβαση ε, στη δουλειά που κάνουν όλοι αυτοί οι σύμβουλοι για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τα οποία χρησιμοποιούν για να κάνουν δουλειέ. Ε, πολλούν αυτές τις πληροφορίες τις οποίες έχουν πρόσβαση στην ΣΥΔΙ του Λονδίνου τις οποίες θα πληρώνουν αδρά. Ναι, εντάξει, αυτό φέρνει χρήματα ε, για το ΑΕΠ της Ευρώπης, αλλά εγώ έχω εντυπωσιαστεί πολύ αρνητικά. Όπως είπατε, δεν έχουμε επόπτες και χρειάστηκε να ε, καλέσουμε εξωτερικούς, αλλά μου κάνει εντύπωση ένας δημόσιο οργανισμός όπως ο δικός σας που ασκεί ε, ε, ένα έργο που υπερασπίζεται τα συμφέροντα της κοινωνίας δεν έχει άλλη επιλογή από το να αναθέσει τη δουλειά της σε μια τέτοια επιχείρηση. Πραγματικά αυτό με οδηγεί να σκεφτώ ότι πρέπει να διακόψουμε τέτοιου είδους εξαρτήσεις. Σε ό,τι αφορά τις διοντολογικούς κανόνες, επειδή οι εθνικοί επόπτες ε, είχαν παρόμοια θέματα να αντιμετωπίσουν και τα εθνικά κοινοβούλια ε, ενδεχομένως επίσης ε, έθεταν ερωτήματα. Θέσαμε υπόψη τους τις, αρχές τις συμφωνίες εμπιστευτικότητας και τους διοντολικούς κανόνες που έγιναν δεκτοί στη συμβάση που υπογράψαμε. Υπάρχουν κανόνες πολύ αυστηροί ό,τι αφορά το χειρισμό των δεδομένων, οπότε πιστεύω ότι κάναμε ό,τι μπορούσαμε προκειμένου όλα να λάβουν χώρα με ηθικό τρόπο στο μέτρο του δυνατού. Τώρα, αν λένε στο City ότι η ΕΚΤ ζητά τον επαναπατρισμό των συναλλαγών ε, στο, στην Ευρωζώνη Ευρώ, ε, δεν καταλαβαίνω γιατί θα τους πιστέψει το City, διότι δεν ζητούμε κάτι τέτοιο. Η ΕΚΤ δεν ζητά κάτι τέτοιο δεν νομίζω θα έπρεπε να αμυφθούν ε, οι σύμβουλοι ε, για τέτοιου είδους συμβουλές. Ε, εμείς ε, λέμε ότι οι υποδομές τους θα πρέπει να είναι στη ζώνη ευρώ, ε, αλλά αυτό είναι κάτι δημόσιο. Δεν είναι κάτι το κρυφό ή το εμπιστευτικό έτσι ώστε να πρέπει κάποιος να πληρωθεί για να τους το πει. Νομίζω ότι οι συνθήκες στις οποίες λαμβάνει η χώρα η, αξιολόγηση είναι ιδιαίτερες. Δεν πρόκειται να έλαβε μάλλον χώρα η αξιολόγηση ε, και εξακολουθεί να λαμβάνει. Ε, είναι ιδιαίτερες διότι δεν είχαμε το παρκές ε, προσωπικό για να κάνουμε την αξιολόγηση μόνοι μας. Εν τω μεταξύ η διάσταση του εγχειρήματο είναι τεράστια. Σας μίλησα για τι νούμερα κάνουμε λόγο. Ακόμα και με τη βοήθεια των εθνικών εποπτών, εποπτικών αρχών, δεν θα μπορούσαμε να το αναλάβουμε χωρίς εξωτερικούς συμβούλους. Οπότε ε, το μη χείρον βέλτιστον. Η, το πανόραμα ήταν πραγματικά πολύ περίπλοκο. Η διακυβέρνηση, οι διαδικασίες της ΕΚΤ σας βεβαιώ ότι είναι άψογες. Αργ, αργοί αργούν, αλλά είναι εξαιρετικές διαδικασίες. Ευχαριστώ πολύ κυρία Νούη. Μπορώ να σας κάνω μια ερώτηση στα ισπανικά, λέει ο πρόεδρος. Ε, μπορείτε να είστε λίγο πιο συγκεκριμένοι σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα ε, των stress test και της, ε, του ελέγχου ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού. Ναι, οι, οι εθνικοί επόπτες και οι τράπεζες θα πρέπει να σεβαστούν το χρονοδιάγραμμα των stress test και του ελέγχου ποιότητας. Ασφαλώς εξ αρχής προβλεπόταν ότι το τέλος ε, του ελέγχου ποιότητας και η αρχή του, των stress test θα αλληλοεπικαλυφθούν λίγο. Ε, έχουμε και το χρονοδιάγραμμα της CBA, οπότε για τον έλεγχο της ποιότητας θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να τελειώσουμε αρκετά νωρί ώστε να ξεκινήσουμε τα stress test. Αυτή τη στιγμή όμω έχουμε τηρήσει το χρονοδιάγραμμα πλήρω. Πρόεδρο, ευχαριστούμε πολύ κυρία Νόη που ήσασταν εδώ μαζί μα για την πρώτη αυτή τακτική δημόσια ακρόαση. Σα υπενθυμίζω ότι η επόμενη ακρόαση θα λάβει χώρα στι 7 Οκτωβρίου. Δεν ξέρω ποιοι θα είναι εδώ. Εσεί θα είστε εδώ κυρία Νόη σίγουρα. Ευχαριστώ. Ε, περιμένω λοιπόν να γνωρίσω τα μέλη της επόμενης ε, σύνθεσης Επιτροπής ε, ΕΚΟΝ. Ευχαριστώ.